πολύ δύσκολη και δυστυχώ έχουμε πολλέ άλλε προτεραιότητε προτού εξαλειφθεί η, η προξενική θεώρηση. Σε μια Ευρώπη που έχει πολλά προβλήματα με την παράνομη μετανάστευση, δεν νομίζω ότι το Συμβούλιο θα δείξει ιδιαίτερο ζήλο για να υπάρξει αυτή η άρση τη ανάγκη προξενική θεώρηση. Είναι λοιπόν κάπω πρόωρο αυτό. Και αναφέρομαι στο τελευταίο κομμάτι της, παρα... της συμβαστικής Τοπολογίας 25. Αυτά. Ναι. Ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Αλμπερτίνη. Πριν από αυτό, ε, θέλω να συμφωνήσω με την πρόταση της κυρίας Ντεκάιζερ. Η πρότασή της μου φαίνεται σωστή και λεπτή. Ε, το λόγο έχει ο κύριος Αλμπερτίνη, ο πρόεδρος, ο πρώτος, ο πρώην πρόεδρος. Όχι, όχι, συνάδελφο, συνάδελφε να με αποκαλείτε. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Θα ήθελα να ε, ανταποδώσω και εγώ στις ευχαριστίες που άκουσα, τις δικές μου ευχαριστίες για όσα ανταλλάξαμε. Δεν είναι πάντα εύκολο να καταλήγει κανείς σε συμβιβασμό ε, και μάλιστα τόσο θετικό. Ε, είναι πάντα δύσκολο να υπεκεραστούν οι δυσκολίες. Μερικές παρατηρήσεις πάνω στα επιχειρήματα που άκουσα. Στο συνάδελφο Ντάφα. Ο κύριος Ντάφα τονίζει όλος ιδιαιτέρως ε, αυτά που συμβαίνουν. Θέλει λίγο να εμφανιστούμε πιο αποφασιστικοί, πιο κατηγορηματικοί στην διατύπωση των ευχών μας. Εμείς θεωρούμε ότι οι όροι που χρησιμοποιήσαμε είναι αυτοί που είναι αποδεκτή στο σημερινό στάδιο των εξελίξεων. Εξελίξεις που δεν είναι επαναστατικές. Έτσι όπως το έχουμε διατυπώσει ε, με μια έντονη επιφυλεκτικότητα προσπαθώντας να καταλήξουμε στην πιο ισορροπημένη διατύπωση που θα μπορέσει να κερδίσει τη συμφωνία του μεγαλύτερου αριθμού των συναδέλφων. Αναφέρω, δεν θέλω να παραθέσω τον Βολτέρο, ε, ε, σέβομαι την άποψη των συναδέλφων, και δεδομένου ότι έχει υποβληθεί και μια έκθεση μειοψηφίας που είναι στον αντίποδα της δικής μας, ασφαλώς δίκιο θα έχει από την πλευρά του, αλλά ωστόσο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, έτσι δεν είναι, εφόσον η δική του είναι έκθεση μειοψηφίας. Προς τον συνάδελφο Τάνοκ, ε, νομίζω πρέπει να δώσουμε κάποιες διευκρινήσεις εδώ, γιατί κάποιες από τις αντιρρήσεις που εξέφρασε ε, έχουν ληφθεί υπόψη στις προφορικές τροπολογίες. Ε, δεν τις είδα γιατί έφτασαν την τελευταία στιγμή. Αναφέρομαι, ο κύριος, η κυρία Ντικάιζερ το ανέφερε εξάλλου για τη σύλληψη του Γκμπάμπο, τροπολογία 3 ή συμβιβαστική τροπολογία 24, όπου γίνεται λόγος για την Ταϊβάν στην πραγματικότητα. Ίσως όχι με την ακρίβεια των όρων που θα ήθελε εκείνος, πάντως αυτά είναι συμβιβαστικές τροπολογίες και προφανώς ε, ε, διατυπώνονται με τρόπο συνθετικό. Η συνάδελφος Λούνατσεκ έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία για την για μια αποκλαστικά πολιτική και όχι στρατιωτική προσέγγιση. Την άποψή της ασφαλώς τη συμμεριζόμαστε, αλλά στην πρότασή της διατυπώνονται και κάποιες, κάποια κριτική για τη θέση του ΝΑΤΟ, ε, στο οποίο όμως ανήκουν ε, τα περισσότερα κράτη που ανήκουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Υπάρχει η υποχρέωση κάποτε να χρησιμοποιηθούν και μέτρα βίας, ε, κατακριτέα συνήθως, αλλά μερικές φορές δεν γίνεται διαφορετικά. Ε, τι θα γινόταν αν είχαμε αντιδράσει όπως ο Γκάντι ε, όταν πριν από 60 χρόνια ο Χίτλερ ήθελε να επιβάλλει το δικό του όραμα για τον κόσμο. Κάποτε είναι απαραίτητη και η βία. προς τον, στην, η συνάδελφος Ντεκάιζερ έγιρε κάποιες αντιρρήσεις για τον όρο που χρησιμοποίησε η κυρία Άστον. Εμείς αναγκαστικά ε, χρειάστηκε να αντιγράψουμε αυτό που λέγεται η υπουργό των εξωτερικών μας σε εισαγωγικά. Ε, ε, βέβαια, μια τροποποίηση της τροπολογίας που μιλάει για το welcomes, χαιρετίζει για κάτι πιο ήπιο, καταγράφει, σημειώνει, δεν ξέρω, notes ή κάτι τέτοιο, μπορούμε σίγουρα να βρούμε μια άλλη διατύπωση. Στη συνέχεια, για την τροπολογία 13, το λεπτό επιχείρημα, το οποίο αφορά την Τουρκία. Και εδώ νομίζω ότι η διατύπωση που υιοθετήσαμε μετά και από την παρέμβαση του συναδέλφου Κασουλίδη και Ντανζάν ε, κάναμε πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό στο πλαίσιο της δικής μου ομάδας και εν πάση περιπτώσει η διατύπωση που χρησιμοποιούμε εκφράζει την σύμπτωση των απόψεων της ανάγκης που υπάρχει να αναγνωρίσει η χώρα αυτή την πλήρη νομιμότητα ε, και την εδαφική ακαιρεότητα μιας χώρας μέλους ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, σε αυτή τη λεπτή φάση που περνάμε, όπου συμμετέχουμε όλοι μαζί στο ΝΑΤΟ και όπου έχουμε και ένα διάλογο με τον ανατολικό κόσμο, ε, χρησιμοποίησαμε μια διατύπωση που μας φαίνεται χρήσιμη. Παραμένει πάντως η αίτηση για χωριστή ψηφοφορία ε, και μπορεί ο καθένας να πάρει θέση ανάλογα με την προτίμησή του. Εγώ ως εισηγητής δέχομαι και συμμερίζομαι κιόλα τις απόψεις αυτές για τη χωριστή ψηφοφορία. Τώρα, ως ομάδα έχουμε αμέσως μετά μια συνεδρίωση και ίσως πριν από την αυριανή ψηφοφορία, ε, αν χρειάζεστε κάτι καινούριο, να απευθυνθείτε και στους κοιόδης εισηγητές και ευχαριστώ για την προσοχή σας, Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια εισηγητά Αλμπερτίνη για το εξαιρετικό έργο. Η ψηφοφορία προβλέπεται για αύριο στις 10, ημέρα Τετάρτη. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Bene, Καλώς. Λοιπόν, μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάτηξης για την ανάπτυξη της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας μετά την έναρξη της ισχύω της συνθήκης της Λισαβόνας. Η Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας, η Υποεπιτροπή, ήδη εξέτασε το Φεβρουάριο αλλά και στις 15 Μαρτίου και, σε τρίτη φάση στις 4 Απριλίου το σχέδιο έκθεσης ε, του κυρίου Γκουαλτιέρη. Α, Νάτος, εντάξει, εδώ είναι, γιατί πριν τον έβλεπα να κάθεται δίπλα στον κύριο Μπρόκ. Εντάξει, εδώ είναι ε, που αφορά ακριβώς τον τίτλο που ανέφερα. Υπάρχουν 284 τροπολογίες. Ο εισηγητής είχε πολλές και στενές επαφές με τους σκιώδεις εισηγητές. Η έκθεση του ε, συνδέεται πολύ στενά με την έκθεση ε, τη δική μου. Η ΚΕΠΑ και η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας είναι πολύ στενά συνδεδεμένες και εξελίσσονται παράλληλα σίγουρα με επικεφαλή στην κυρία Άστον και άλλους αρμόδιους. Ε, δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Ε, ευθύς εξ αρχής να συγχαρώ τον εισηγητή ε, Γκουαλτιέρη για όλο το έργο που έφερε σε πέρας και ε, αναμένω να ακούσω τα σχόλιά του. Του δίνω το λόγο λοιπόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, δεν θα μπω σε αναλυτική παρουσίαση της έκθεσης, γιατί ήδη την έχουμε συζητήσει εκτενώς στην Υποεπιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας. Ωστόσο κάτι θα πω ε, επί της ουσίας και επί των κυριότερων σημείων ε, της εργασίας που μας επέτρεψε να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες οι οποίες αντανακλούν τη συνένεση και τη συμφωνία της πλειοψηφίας των πολιτικών ομάδων. Και έχουν υποβληθεί και προφορικές τροπολογίες, οι οποίες ε, τροποντινά μας επέτρεψαν όπως ακριβώς συνέβη και με τη δική σας εισήγηση κύριε Πρόεδρε, να επικαιροποιήσουμε την έκθεση εν ώψη και των πρόσφατων εξελίξεων. Το θέμα της έκθεσης αυτής ήταν η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας υπό το φως της συνθήκης της ε, Λισαβόνας και προσθέτω και εν ώψη των εξελίξεων του διεθνού συστήματος. Και προσπάθησα να εμείνω πιστός στο καθήκον αυτό για να επιτευχθεί και μια συμπληρωματικότητα μεταξύ της σχέσης ε, της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και της πολιτικής ΚΕΠΑ. Δεν ξέρω κατά πόσο δεν έχετε... οι συνάδελφοι που δεν συμμετείχαν στις συζητήσεις στην Επιτροπή Άμυνας και Ασφάλειας θα δούνε τους γενικούς πολιτισμούς της κοινή εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στους διάφορους διεθνείς ε, παίκτες. Μία από τις βασικές θέσεις της έκθεσής μου είναι ότι πρέπει να υπάρξει πολύ στενή ε, μια πολύ στενή να υπαρξει πολυ μια μεταξύ της ΚΕΠΑ και της ΕΠΑ. Ε, να υπάρξει μια συγκεντρωτική, ολοκληρωμένη, ενιαία προσέγγιση. Εγώ λοιπόν έμεινα στην ουσία ότι θεώρησα ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η ολοκληρωμένη ενιαία προσέγγιση στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας στην Ευρώπη έτσι ώστε να ανταποκρινόμαστε στις εξελίξεις του διεθνούς σκηνικού. Να μην υπάρχει ε, μια μονόπλευρη προσέγγιση που θέλει την Ευρώπη ως μόνη και κυρίαρχη, ε, ως Ευρώπη και έτσι μέσα στη σημασία της, αλλά να αναγνωρίζει την αλληλεμένων που καθιστούν την άμυνα ένα πολυδιάστατο ε, φαινόμενο. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια σφαιρική προσέγγιση. Δεν μπορούν να εξετάζονται κατηδίαν τα θέματα της ασφάλειας, της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί η ασφάλεια επισέρχεται παντού, στις ε, σχέσεις, στις επιχειρήσεις, στην εξωτερική πολιτική. Ε, σε όλα τα κεφάλαια της έκθεσής μου. Δεν μπορεί λοιπόν να αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστό θέμα. Ο κίνδυνος που υπήρχε στο παρελθόν λόγω της ε, αδυναμίας της ε, πολιτικής εξωτερικής πολιτικής υπήρχαν επιχειρήσεις που διεξάγαμε, αποτελεσματικές κιόλας, αλλά επειδή ακριβώς δεν εντάσσονταν σε μια συνολική στρατηγική εξωτερικής πολιτικής, εν τέλει δεν ήταν όσο αποτελεσματικές όσο θα μπορούσαν να είναι. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι και το μέγεθος της έκθεσης και το γεγονός ότι δεν αναπτύσσονται πολύ σχέσεις με τη Ρωσία, την Κίνα, τη Μέση Ανατολή. αυτό το έκανα ακριβώς για να υπάρχει αυτή η στενή σύνδεση που ανέφερα μεταξύ της εξωτερικής πολιτικής και της κοινή πολιτικής άμυνας και ασφάλειας. Αυτή η αναγκαιότητα για μια σφαιρική προσέγγιση δεν απορρέει μόνο από, το, από την φύση του κόσμου ως εν, ενός κόσμου πολλαπλών πόλων. Αλλά η σφαιρική αυτή προσέγγιση μας επιτρέπει να επιτύχουμε και πολύ περισσότερα από όσα έχουμε επιτύχει στο παρελθόν. Και αυτό είναι ένας από τους σκοπούς της έκθεσης, να δούμε πώς και κατά πόσο η συνθήκη της Λισαβόνας, με τη σωστή της ερμηνεία, μπορεί να μας ε, βοηθήσει να ενισχύσουμε αυτή την αντίληψη για την ασφάλεια ως στοιχείο που εντάσσεται σε μια γενικότερη προσέγγιση. Χωρίς να επισέλθω στην ουσία του περιεχόμενου της έκθεσης, όλα γραπτά είναι, έχω τη γνώμη ότι η συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, εναρμονίζεται πλήρως με αυτήν την απέτηση μιας σφαιρικής προσέγγισης και μας παρέχει εργαλεία σε επίπεδο δομικό, οργανικό, αρχιτεκτονικό, ε, αλλά μας δίνει και νομικά μέσα επίσης να εντάξουμε σε ένα ενιαίο σύνολο την κοινή εξωτερική πολιτική και την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό βέβαια προϋποθέτει μια σειρά από πολιτικούς όρους, ε, κάποια θεσμικά, νομικά μέσα. Αλλά εγώ φυσικά στην έκθεσή μου και στις προφυρικές τροπολογίες περιορίστηκα ε, να τονίσω κάτι που δεν μπορούμε να αγνοούμε και συγκεκριμένα ότι απέναντι στις κύριες στρατιωτικές επιχειρήσεις των τελευταίων χρόνων η Ευρώπη έλαβε μέρος. Ε, ο κύριος Αλμπερτίνη έχει ασχοληθεί πιο εκτενώς με το θέμα αυτό, αλλά εγώ από την πλευρά μου ήθελα να τονίσω ότι δεν είναι δυνατόν να θεωρούμε την κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας ως κάτι που στο οποίο συμμετέχει ένα ευρωπαϊκό κράτος μέλος μόνο και μόνο επειδή είναι ευρωπαϊκό κράτος. η, πολιτική, η κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας τελικά εξαντλείται σε κάποιες δράσεις που διεξάγουν ορισμένα κράτη-μέλη επειδή έτυχε να συμφωνήσουν. Ε, δεν μου αρέσει αυτή η ερμηνεία και νομίζω ότι πρέπει να εγκαταληφθεί αυτή η προσέγγιση. Αντιθέτως πρέπει να αξιοποιηθούν τα μέσα που μας παρέχει η συνθήκη ακόμα και αν παραχωρηθεί σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη να διεξάγουν επιχειρήσεις κοινή ευρωπαϊκής πολιτικής άμυνας και ασφάλειας, ε, ακόμα και αυτό είναι βέβαια δυνατόν. Ε, μας το επιτρέπει η συνθήκη της Λισαβόνας, αλλά αυτό πρέπει να βασίζεται σε απόφαση του Συμβουλίου που θα ορίζει τα όρια της σχετικής δράσης και το περιεχόμενό της ε, σε συμφωνία και με τα άλλα όργανα. Ακόμα και υπό αυτήν τη μορφή. Η συνθήκη της Λισαβόνας μας το επιτρέπει. Και νομίζω ότι έτσι μπορούμε να διατηρήσουμε και την τάξη μεταξύ μας και να μην υπάρχουν διαφωνίες και διασπαστικές τάσεις. Λοιπόν, χωρίς να μπω στα διάφορα κεφάλια ε, της έκθεσής μου, θα ήθελα να αναφέρω ε, την αναζήτηση ενός συμβιβασμού για τον ρόλο της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, η οποία όπως διαμορφώθηκε στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων είναι ακριβώς ένας θεσμός που θα ασχολείται με την ε, γενική, με τη σφαιρική εξωτερική δράση ε, θα έχει και θα έχει ως αντικείμενο και την παροχή βοήθειας προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο με στόχο την ανάπτυξη και στρατιωτικές δράσεις. Θα είναι ένα είδος υπηρεσίας διαχείρισης κρίσεων. Ε, ε, έτσι ακριβώς αναδύθηκε από τις διαπραγματεύσεις. Και έτσι και εγώ την ε, σκέφτηκα να μην νομιστεί ότι θέλουμε να ιδρύσουμε μια καινού, ένα καινούργιο όργανο, μια καινούργια υπηρεσία που θα διαταράξει τα νερά και τις σχέσεις μας με τον ύπατο αρμοστή και με τον ύπατο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 είναι λοιπόν μία μονάδα ε, η οποία θα συνεδριάζει τακτικά και θα μπορεί να εκπονεί κάποια σχέδια, κάποια προγράμματα και να ορίζει ε, μορφές διαχείρισης των κρίσεων ε, έτσι ώστε η Ευρώπη να μπορεί να χρησιμοποιεί τα διάφορα μέσα που έχει στη διάθεσή της με συνακτικό και ευφυή τρόπο. Είμαι υπέρ λοιπόν τη συμβιβαστική λύση στην οποία καταλήξαμε και ευχαριστώ τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες για τη βοήθειά τους. Τώρα, ως προς τα πιο ζωτικά σημεία της έκθεσης. Ε, σας αναγγέλω ότι θα προτείνω, σας ανακοινώνω ότι θα προτείνω άλλη μια προφορική τροπολογία, μάλλον μία μόνο είναι ούτως ή άλλως, για την πρότασή μου για τις battle group, για τις μάχημες ομάδες κατανοώ ότι η διατύπωση έτσι όπως την έχω εντάξει, να υπάρχει μια μάχημη ομάδα και μια υποδεέστερη μάχημη ομάδα και έτσι όπως περιγράφω τους τύπους των επιχειρήσεων, είναι μια πρόταση αρκετά αναλυτική ίσως, να διατηρήσουμε μόνο το πολιτικό μήνυμα αυτής της πρότασης. Θα προτείνω λοιπόν μια προφορική ορολογία η οποία δεν θα λέει should be κτλ. κτλ αλλά να πω ότι μπορεί να εξεταστεί και το ενδεχόμενο χρήσης κτλ. Μια πιο ήπια διατύπωση λοιπόν, έτσι ώστε να καταστεί αποδεκτή από όλες τις ομάδες. Γιατί νομίζω ότι και το Κοινοβούλιο μπορεί να συμβάλλει και από αυτήν την άποψη. Δίπλα στην άλλη εκείνη πρόταση, η οποία μου φαίνεται πολύ λογική και στην οποία συμφώνησαν και οι άλλες πολιτικές ομάδες, να καλυφθεί το κόστος αυτών των μάχημων ομάδων ε, από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 το να υπάρχει μια αποτελεσματική αγορά άμυνας στην Ευρώπη, χωρίς την οποία δεν έχει νόημα η αναρδιάρθρωση της, ε, ε, του κλάδου και των βιομηχανιών άμυνας και ασφάλειας. Πρέπει να, ο κλάδος αυτός να είναι ανταγωνιστικός στο σημερινό κόσμο, να υπάρξει καινοτομία, να υπάρχει ανάπτυξη στον τομέα αυτό της άμυνας. Ε, άλλο σημείο η σχέση μεταξύ εξωτερικής και εσωτερικής ασφάλειας, ζήτημα κρίσιμης σημασίας. Κάνω κάποιες προτάσεις, κάποιες συστάσεις, οι οποίες πηγαίνουν προς την κατεύθυνση όσων γίνονται ήδη. Υπάρχει και κοινή εργασία κόψ και κόζι και απαντώντας ε, στην πρόταση της επικεφαλής της υπηρεσίας ε, της αντιτρομοκρατικής της Ευρώπης, να προτείνουμε και αντιτρομοκρατικές δράσεις στο πλαίσιο της Frontex και όλων των άλλων μονάδων που δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή εκφράζοντας την Ευρώπη. Δεν ξέρω, ίσως μετά την ψηφοφορία θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Να, λέγαμε κάτι και γι' αυτό. Τέλος, φυσικά, έχοντας ε, συμμετάσχει ως διαπραγματευτής, δεν μπορώ παρά να αναφέρω την ε, ατυχή έκβαση των ε, διαπραγματεύσεων της διακοινοβουλευτικής συζήτησης για την άμυνα και την ασφάλεια και Έχω συντάξει και μια προφορική τροπολογία για, για αυτό και επαναλαμβάνουμε τις θέσεις εκεί του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τέλος ε, υπάρχει και ένα τμήμα της έκθεσης για τις εταιρικές σχέσεις. Με... Πάνω σε αυτό δεν υπάρχουν ιδιαίτερα πολιτικά προβλήματα και επομένως μπορώ να μην μπω αναλυτικά, να σας παραπέμψω στις προφορικές τροπολογίες, στις συμβιβαστικές τροπολογίες και στις τροπολογίες που υπέβαλαν όλοι οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για αυτή την εξαντλητική παρουσίαση. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Ας ξεκινήσουμε από τον συνάδελφο Λίζεκ. Ε, ε, Κυρίες και κύριοι, κατανοώ πολύ καλά ότι ο εισηγητής έχει το δικαίωμα βέβαια να, μιλεί, να μιλήσει όσο θέλει. Ε, αλλά εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι πιο σύντομος κανείς όταν παίρνει το λόγο. Εν πάση περιπτώσει, συμβιβάζομαι. Ξέρουμε ότι η πολιτική της, ε, η κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας είναι ένα θέμα για το οποίο θα μπορούσαμε να μιλάμε όλες ώρες ολόκληρες. Ξέρουμε επίσης ε, ποια είναι τα προβλήματα που έχουμε μπροστά μας. Γνωρίζουμε τα διάφορα προβλήματα που παραμένουν ανεπίλητα λόγω της θέσεως ορισμένων κρατών μελών και ξέρουμε επίσης ότι οι ε, ε, ευρωπαϊκοί θεσμοί ε, βρίσκονται σε εμβριακό στάδιο σε ό,τι αφορά αυτά τα θέματα. Πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ για να βελτιωθεί η συνεργασία. Πιστεύω όμως ότι οι θεσμοί, ο υπατός εκπρόσωπος, ότι ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Άμυνας και όλοι οι άλλοι θεσμοί θα φτάσουν σε ένα ικανό επίπεδο και θα περατώσουν το έργο τους. Το Κοινοβούλιο δεν λαμβάνει αποφάσεις, ε, δεν έχει τη δυνατότητα την πλήρη λήψη αποφάσεων εδώ, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικός ο ρόλος του και αυτό αυτό μας το λένε όλοι όσοι συνεργάζονται με τη Βαρόνια Άστον. Αυτό μας το είπε και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Άμυνας αλλά και όλοι όσοι ασχολούνται με τον ε, τομέα που καλύπτει η έκθεση του κυρίου Γκουαλτιέρη. Η έκθεση είναι πολύ θετική. είναι τόσο ε, θετική που έχει 284 τροπολογίες κατατεθειμένες. Και ο κύριος Γκουαλτιέρη ελπίζω πως θα συμφωνήσει ότι η δική μου πολιτική ομάδα δεν κατέθεσε τροπολογίες που αλλάζουν πάρα πολύ την ουσία. Απλώς εμπλουτίνουν και τελειοποιούν τον λόγο του κατά κάποιον τρόπο. Είμαι απόλυτα ε, ευγνώμων προς τον κύριο Γκουαλτιέρη για τον ανοιχτό χαρακτήρα της σκέψης του, για την ε, ε, βούληση και τη θετική αντιμετώπιση που έδειξε σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες της ομάδας μου. Είχαμε μια πάρα πολύ αγαστή συνεργασία στη συνεδρίαση που είχαμε. Είχαμε θετικές συζητήσεις και η πολιτική μου ομάδα και εγώ επιβεβαιώνουμε ότι θα υποστηρίξουμε όλες τις συμβαστικές τροπολογίες και τις προφορικές τροπολογίες. Ευχαριστώ κυρία Λίζεκ. Ο κύριος Ντάφα. Ε, um, Πρόεδρε, έχουμε εδώ μία εξαιρετικά ουσιαστική και εμπεριστατωμένη έκθεση για την, για την πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Είναι πραγματικά εμπεριστατωμένη λόγω της εμπειρίας του κυρίου Γκουαλτιέρη, ο οποίος υπήρξε και ένας από τους δύο διαπραγματευτές μας για την ε, ίδρυση <clears throat> της ε, υπηρεσίας εξωτερικής δράσης. Που είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη και ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο δρόμο της ανάπτυξης της διάστασης ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι είναι μια καλή έκθεση, γιατί δεν αντιμετωπίζει με χαλαρό τρόπο τα προβλήματα αυτά, έχει πιο επικριτικό και κριτικό πνεύμα από τις προηγούμενες εκθέσεις μας για τα θέματα αυτά, εν μέρει διότι έχει εφαρμοστεί ήδη η συνθήκη της Λισαβόνας και είναι ορθό και πρέπει να ασκήσουμε πίεση για να έχουμε περισσότερα αποτελέσματα το αν ε, αν εκφράζει λύπη ή εκφράζει βαθιά λύπη για το ψήφισμα 1973 του Συμβουλίου Ασφαλείας, αυτό είναι μια συζήτηση η οποία μπορεί να συνεχίσει στο Δινεκές. Εγώ κατανοώ αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κασουλίδης για τις ιδιαίτερες ευαισθησίες που μπορεί να έχει η Γερμανία στο να συμμετέχει σε στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αλλά και εμείς έχουμε κάθε δικαίωμα να πούμε ότι θέλουμε η Γερμανία να έχει περισσότερη αυτεπίγνωση ως συμμετέχον, ως εταίρος στην ανάπτυξη της ΕΠΑ και είναι κρίμα που κάποια κράτη-μέλη και κυρίως αυτό αναφέρεται στην ε, Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν χρησιμοποίησαν τις πρόνοιες της συνθήκης για να αναπτύξουν ειδικέ αποστολές εξ της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. και ουσιαστικά έφεραν σε πέρα στην ίδια αποστολή σε ένα πλαίσιο που ήταν εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως κοινοβουλευτικοί λοιπόν εμείς που είμαστε υπεύθυνοι για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο της άσκησης της ε, κοινή εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, ιδίως στον τομέα της ΕΠΑΑ, νομίζω ότι είναι πολύ σωστό να εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας και να προσπαθήσουμε να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν περαιτέρω τη συνεργασία στον τομέα της ε, ΕΠΑΑ όπως προβλέπει και η συνθήκη, ώστε να υπάρξει πλήρης ανάπτυξη των ε, διατάξεων της ε, συνθήκης που έχουν σμιλευτεί με μεγάλη τέχνη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ακριβώς σενάρια όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε σήμερα στη Λιβύη. Και επομένως η συμβαστική τροπολογία 6 πιστεύω ότι θα είναι απαραίτητη η σωστή διατύπωση της αντίδρασής μας στην ε, επιθετική συμφωνία μεταξύ των ε, Βρετανών και των Άγγλων. Να επιλέξουμε λοιπόν πολύ προσεκτικά τα λόγια μας. Μπορούμε να εκφράσουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι αυτή η επιχείρηση δεν έλαβε χώρα μέσα στα πλαίσια της συνδίκης Λισαβόνης. Μπορούμε όμως να δώσουμε και μία αισιόδοξη νότα στο γεγονός, τονίζοντας το γεγονός ότι έγινε αυτή η επιχείρηση παρόλα αυτά, και ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν και περαιτέρω βήματα στη συνεργασία στον αμυντικό και ασφαλίτικο τομέα. Θα ήθελα να επαναλάβω αυτά που είπα σε σχέση με την έκθεση του κυρίου Αλμπερτίνη. Είναι μια έκθεση που θα πρέπει να δημοσιευθεί και να τύχει πρόθεσης προς τα Εθνικά Κοινοβούλια γιατί είναι σαφές πλέον από την πρόσφατη αποτυχία να υπάρξει συμφωνία με τα Εθνικά Κοινοβούλια για μια κοινή προσέγγιση στα θέματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου της ΕΠΑ καθώς και της ΚΕΠΑ. Είναι φανερό λοιπόν από όλα αυτά ότι υπάρχει ακόμα η εντύπωση στα Εθνικά Κοινοβούλια ότι όλα αυτά τα οποία εμπίπτουν στην πολιτική άμυνας και ασφάλειας πρέπει να παραμείνουν σε ένα επίπεδο διακυβερνητικής άσκησης. Αποκλείοντας λοιπόν οτιδήποτε δεν ενδιαφέρει τις εθνικές κυβερνήσεις και θεωρούν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να συμμετέχει στον κοινοβουλευτικό έλεγχο αυτής της πολιτικής και αντίθετα θα πρέπει να περιοριστεί στον ρόλο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης η οποία μπορεί να συζητά και να κρίνει τα θέματα της ήπιας ασφάλειας και της ήπιας άμυνας. Εμείς λοιπόν δεν πρέπει να δεχτούμε μια τέτοια αντιμετώπιση, θα πρέπει να αρνηθούμε να συμπλέψουμε με την πρόταση πολλών εθνικών κοινοβουλίων που θα ανοίγαγε το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο να είμαστε απλώς και μόνο στα επίπεδα, σε ένα ελάχιστο, σε ένα παράλογο επίπεδο, κάτι το οποίο δεν φύγει μονάχα το κύρος και την αξιοπιστία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά εξάλλου δεν λαμβάνει και υπόψη και δεν σέβεται την λογική της συνθήκης της Λισαβόνας και εξάλλου θα αποδυναμώσει και την ικανότητα να υπάρξει μια κοινοβουλευτική απάντηση στην ανάπτυξη και παρακολούθηση στην ανάπτυξη της ΚΕΠΑ και ΕΠΑ. Αυτά που λέγονται λοιπόν στη συμβαστική τροπολογία C, κατά την απόψή μου, είναι απόλυτα ορθή η διατύπωση αυτή. Θα πρέπει με ευγένεια να εκφράσουμε τη λύπη μας για το γεγονός ότι δεν υπήρξαν οι απαραίτητες διαπραγματεύσεις και δεν καρποφόρησαν οι διαπραγματεύσεις με τα Εθνικά Κοινοβούλια, θα μπορούμε να είμαστε υπομονετικοί, να περιμένουμε να έρθουν καλύτερες μέρες και να λειτουργήσουμε μέσω των κομματικών δικτύων μας για να προσπαθήσουμε να μεταπίσουμε τους εθνικούς συναδέλφους μας και να υπάρξει καλύτερη κατανόηση στα Εθνικά Κοινοβούλια του κομβικού ρόλου που θα πρέπει να διαδραματίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να παρακολουθήσει, να ελέγξει και να διαρθρώσει τα κοινά στοιχεία στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Η ομάδα μου λοιπόν θεωρεί ότι η έκθεση Γουαλτιέρη είναι ένα σημαντικό βήμα προς το εμπρός για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε την ε, ανάδυση μια αμοιβαία κατανόηση μεταξύ ημών και των Εθνικών Κοινοβουλίων. Ευχαριστώ κύριε Ντάφα. Ο κύριος Τάνοκ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Τα σχόλιά μου θα είναι σύντομα γιατί ε, υπάρχουν μια σειρά από ε, τροπολογίες κλειδιά που έχουν υποβληθεί στην έκθεση. Θα ήθελα να πω ότι ε, είναι ένα μακροσκελές κείμενο με 80 παραγράφους και με 240 ε, τροπολογίες. Νομίζω ότι πρέπει να δούμε τις διάφορες ρυθμίσεις σχετικά με την άμυνα, με τη διακυβερνητική συνεργασία των ΝΑΤΟ. Ε, εδώ ε, ε, έχουμε ορισμένες επιφυλάξεις για την πολιτική άμυνας αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε υπέρ των διαφόρων επιχειρήσεων όπως είναι η Αταλάντη στην Βόρεια Αφρική τις οποίες υποστηρίζουμε Αταλάντα με συγχωρείτε ε, σε, σε ένα ορισμένο σημείο υπάρχουν ορισμένες ρυθμίσεις ε, βρετανογαλλικές ε, στην Μπαγκόκ υπάρχει προστασία του άμαχου πληθυσμού και κατά κάποιο τρόπο βλέπουμε ότι είναι πάρα πολύ ε, σημαντική αυτή η δραστηριότητα. Δύο χρόνια πριν περίπου είχαμε γνωρίσει αυτή την πολύ ένδοξη περίοδο και υπήρχε ένας αποκλεισμός μας από το θέατρο των επιχειρήσεων στη Νότια Μεσόγειο. Ε, στην περίπτωση της Λιβύης ε, πήραμε όμως ένα ε, ρόλο και υπάρχουν πάρα πολλές τροπολογίες οι οποίες έχουν διαγραφεί και υπάρχει μια ανεπάρκεια σε ό,τι αφορά τις τροπολογίες που αφορούν την πολιτική της άμυνας. Νομίζω ότι η πολιτική της άμυνας είναι ένα πρωταρχικό σχέδιο για τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Λόζινγκ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρία Γκουαλτιέρη, Ήδη στο Στρασβούργο στη συνεδρίασή μας είχατε αναφέρει ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα μιας συμβιβαστικής τροπολογίας με την ΚΟΕ, η οποία τελικά όμως δεν καρποφόρησε και καταλαβαίνουμε απόλυτα την στάση σας σε σχέση με την κοινή εξωτερική πολιτική, πολιτική ασφάλειας, καθώς και την πολιτική άμυνας και ασφάλειας. Και κατανοώ αυτά τα οποία θέλετε να πείτε. Βέβαια, θεωρώ λυπηρό ότι ιδίω στην προφορική τροπολογία 16-ΝΕΑ εσείς έχετε παρουσιάσει την εικόνα μιας ακόμα πιο ενισχυμένα παρεμβαίνουσας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέτε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να παίξει το ρόλο του διαμεσολαβητή και του εγγυητή της ειρήνης. Αυτό το χαιρετίζω. Το να μπορέσει η Ευρώπη να είναι ένας μεσολαβητής είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Αλλά όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, ο ρόλος αυτός ο μεσολαβητικός δεν μπορεί να στέφεται από αξιοπιστία. Πολύ πιο εύκολο θα ήταν η Ευρώπη να περιοριστεί σε πολιτικά και διπλωματικά μονάχα μέτρα. Η προφορική σας τροπολογία επίσης ε, στο σημείο 13 για τον έλεγχο της ΚΕΠΑ και της ΕΠΑ, εδώ υπάρχει μεγαλύτερη σημασία που πρέπει να δοθεί σε αυτό τον έλεγχο, αλλά δεν δίνεται συγχρόνως κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις για την βελτίωση του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Αυτό είναι λυπηρό, γιατί ήδη υπάρχουν πολλές προτάσεις οι οποίες συζητούνται από τα κράτη-μέλη, που δεν λαμβάνουν υπόψη. Επίσης, αναφέρεστε στη συμπερίληψη ορισμένων πολιτικών τομέων όπως είναι η ανάπτυξη και η εμπορική πολιτική στα πλαίσια της κοινή πολιτικής ασφάλειας. Επίσης ζητάτε την αύξηση της συνεργασίας του πολιτικού με το στρατιωτικό τομέα, κάτι το οποίο γνωρίζω ότι πολλοί συνάδελφοι το θέλουν. Και επίσης υπάρχει μια σειρά από πολλαπλές αναφορές στην ε, στρατιωτική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι οδηγεί σε μεγαλύτερη σταθερότητα στο παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης, δεν νομίζω ότι οι τροπολογίες σας μπορούν να αντιμετωπίσουν τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η σταθερότητα και η ειρήνη στον κόσμο μας. Όπως είπε και ο κ. Μάιερ προηγουμένως, για την έκθεση Αλμπερτίνη εμείς θα απορρίψουμε συνολικά την έκθεσή σας και θα καταθέσουμε μια έκθεση μειοψηφίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λόζινγκ. Και τώρα ας δώσουμε τον ε, λόγο στον εισηγητή για τα τελικά του σχόλια. Κύριε Γκουαλτιέρη, έχετε το λόγο. Ε, δεν έχω και πολλά να προσθέσω στην πραγματικότητα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ε, πολιτικές ομάδες για την επικοδομητική συμβολή τους. Πραγματικά ε, θεωρώ το μεγάλο ρυθμό τροπολογιών ε, κάτι το θετικό, γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις επρόκειτο για τροπολογίες που επέτρεψαν ή θα μας επιτρέψουν να εμπλουτίσουμε την έκθεση. Ε, άλλες πάλι τροπολογίες με συνεκτικό τρόπο διαγράφουν μια διαφορετική οπτική ε, ε, οι τροπολογίες της ΓΚΟΕ, οι τροπολογίες του ΕΛΚ. Ε, Συγγνώμη, όχι το ΕΛΚ, το κόμμα των συντηρητικών και των μεταρρυθμιστών. Και σε αυτή την περίπτωση ευχαριστώ τους συνοδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες γιατί και η αρετή του κοινοβουλίου αυτού είναι να μπορεί με πολιτισμένο τρόπο να συγκεράζει διαφορετικές οπτικές. Μία κάτι που είναι αμοιβαία επικοδομητικό και διδακτικό και γόνιμο για την δημοκρατική συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να επαναλάβω για άλλη μια φορά, ε, με κάθε σεβασμό και κάθε κατανόηση της βάσης των θέσεων ε, αυτού του διαρθρωτικού δομικού σκεπτικισμού αν θέλετε, ιδίω από την πλευρά των συντηρητικών και των μεταρρυθμιστών και από την άλλη πλευρά τη ριζοσπαστική οπτική, τη, ριζοσπα... τη ριζική αντίθεση στην χρησιμοποίηση τη βία σε οποιαδήποτε μορφή τη, ακόμα και όταν αυτό μπορεί να γίνει στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και με στόχο την εγγύηση της ειρήνης. Κατανοώ και σέβομαι αυτές τις δύο θέσεις. Φυσικά όμως δεν τη συμμερίζομαι. Και σε αυτή την περίπτωση δεν θα καταφέρουμε να ε, επιτύχουμε σύγκληση απόψεων. Στην περίπτωση των άλλων ομάδων, του ΕΛΚ, ε, των Πρασίνων και των ε, Φιλελεύθερων, θα επέλθει συμφωνία, δεν θα επέλθει συμφωνία και θα καταλήξουμε σε αποκλίνουσες θέσεις ίσως αποκλήσεις πάνω σε μεμονωμένες τροπολογίες. Τροπολογίες ενδεχομένως και σε περιθωριακά ζητήματα. Γι' αυτό και συνολικά ε, θα είμαι πολύ ευτυχής εάν, όπως δείχνουν τα πράγματα, η έκθεση αυτή τελικά θα λάβει τη μορφή ε, καρπού κοινή εργασίας, με θεμητές αποκλήσεις όπως είπα ε, και με κατανόηση από πλευράς μου των ε, αντιρρήσεων που έχουν ε, ορισμένες πλευρές για την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας και την ΚΕΠΑ. Ελπίζω λοιπόν αύριο να ψηφίσουμε ε, κατά συνέπεια των συζητήσεων που είχαμε και νωρίτερα και σήμερα. Ε, Πρόεδρος, ευχαριστώ. Όπως ξέρετε όλοι, η ψηφοφορία για την έκθεση αυτή καθώς και για την προηγούμενη θα, λάβουν χώρα, θα λάβει χώρα αύριο. Θα έχουμε στη διάθεσή μας 7 λεπτά για να αλλάξει η φρουρά και να προετοιμαστεί η επόμενη συνεδρίαση ε, στην οποία θα προεδρεύσει ο κύριος Νίμπλερ, η κυρία Νίμπλερ. Συνάδελφοι, καθίστε στις θέσεις σας παρακαλώ να ξεκινήσουν οι εργασίες της Επιτροπής μας. Η κυρία Νίμπλερ, πρόεδρος της Αντιπροσωπείας, ε, ε, μας είπε ότι ε, συμμετέχει σε κάποια άλλη συνεδρίαση, αλλά θα έρθει. Ωστόσο, μας επέτρεψε να ξεκινήσουμε χωρίς την παρουσία της. Και φυσικά όταν έρθει θα της δώσουμε ε, το χρόνο που της ε, ταιριάζει, που της αναλογεί. Ε, έχουμε μια αντιπροσωπεία που προεδρέπεται από τον κύριο Γιασίμ Αλκαράφη τον ε, χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Όπως ξέρετε στην περιοχή αυτή, ο τίτλος της ε, συνάντησής μας είναι «Ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα σημερινά δημοκρατικά κινήματα στην Αραβική Χερσόνησο, προοπτικές και αντίκτυπο στην περιοχή». Α, έφτασε η συνάδελφος Νίμπλερ. Τι ωραία. Την ευχαριστούμε για την παρουσία της. Στην περιοχή αυτή ε, αναδύονται σημαντικές λαϊκές εξεργές, εξεγέρσεις, ιδίως στο Μπαχρένιν και στην Ιεμένη και, και βίαιη καταστολή η οποία βεβαίως προκαλεί την αποδοκιμασία όλων μας. Προσανα... Προσανατολιζόμαστε προς την απερίφραστη στήριξη των θεμητών προσδοκιών αυτών των λαών για την δημοκρατία και την ελευθερία. Η Επιτροπή μας και η Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο υπό την ηγεσία του συναδέλφου, της συναδέλφου Νίμπλερ και την Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων παρακολουθούν στενά αυτή την κατάσταση. Υπενθυμίζω ότι και ο Αντιπρόεδρος Μπαουντής, Μποντής ε, υπεύθυνο για τις σχέσεις, ε, ε, για τις σχέσεις μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτής της περιοχής του κόσμου. Στην ολο... Εγκρίθηκε το κείμενο κατά την Ολομέλεια της 24ης Μαρτίου. Υιοθετήθηκε επίσης και ένα ψήφισμα, ένα έκτακτο ψήφισμα για την κατάσταση στην Ιεμένη και στο Μπαχρέιν. Ας καλωσορίσουμε λοιπόν και ας ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και προσοχή την παρουσίαση του καθηγητή Φαζ Γκέργκες, του φιλοξενούμενού μας, αναγνωρισμένου ειδικού. Ε, προέρχεται από το London School of Economics και είναι και διευθυντής του Κέντρου για τη Μέση Ανατολή. Σας ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Ε, σας έχουμε ε, διαθέσει ένα περιορισμένο χρόνο για την παρουσίασή σας. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσετε να τον εκμεταλλευτείτε χωρίς να πληγεί από αυτό η σύνθεση των ε, επιχειρημάτων σας και η ακεραιότητα της παρουσίασής σας. 15 λεπτά λοιπόν, έτσι ώστε να δοθεί και χρόνος. Ε, εντάξει, και αν φτάσετε και στα 20 λεπτά ε, εντάξει, αλλά θα σας παρακαλέσω να τηρήσετε τους ε, χρόνους, ε, το χρόνο που σας δίνουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας. Έχω μεταξύ 15 και 20 λεπτά λοιπόν και αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι να παρουσιάσω απλώς μερικές ιδέες και η ελπίδα μου είναι να έχουμε μία ενδιαφέρουσα και καρποφόρα συζήτηση μετά στην ανταλλαγή ερωτήσεων και απαντήσεων. Θέλω να ξεκινήσω κάνοντα μια διευκρίνηση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλη ρευστότητα και αβεβαιότητα στην περιοχή. Όλα αυτά τα οποία σας λέω σήμερα, επομένως, βασίζονται σε μια κατάσταση η οποία είναι ρευστή και εξελίσσεται με μεγάλη ταχύτητα σε όλη αυτή την περιοχή. Αυτό το οποίο βλέπουμε στη Μέση Ανατολή, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο στον Περσικό κόλπο, είναι αυτό που λέω μια εντογενάστε επανάσταση και βρισκόμαστε στην αρχή και όχι στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Τα πράγματα εξελίσσονται με μεγάλη ταχύτητα σε όλη αυτή την περιοχή. Και πιστεύω ότι θα πρέπει να δούμε, να περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η μορφή της Μέσης Ανατολής που θα προκύψει μετά από τις εξελίξεις αυτές. Αυτό το οποίο έχουμε υποτιμήσει ως ερευνητές και μελετητές, ακόμα και πολιτικοί στην ε, περιοχή του αραβικού κόσμου, είναι η δυνατότητα αυτόνομης δράσης. Ξέρουμε ότι υπήρχε μια δομική κρίση, μια κοινωνική κρίση, μια πολιτική κρίση, μια κρίση κυβέρνηση στον αραβικό κόσμο. Αλλά οι περισσότεροι από εμά δεχόμασταν την ιδέα ότι ο Άραβας είναι υποταγμένος, ότι υπάρχει ο παράγον του φόβου, ότι οι αστυνομικές ε, αρχές και το αστυνομικό κράτος θα εμπόδιζαν τους πολίτες από το να αυτονομηθούν και να εξεγερθούν. Και αυτό που είδαμε στους τελευταίους τρεις-τέσσερις μήνες είναι ότι έχει σπάσει το φράγμα του φόβου. Ξέρω ότι αυτό είναι πια ένα κλισέ και η αυτόνομη δράση των Αράβων έχει έρθει στο προσκήνιο. Δεν πιστεύω λοιπόν θα μπορέσει να υπάρξει καμία επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση. Έχει λοιπόν αλλάξει πραγματικά η κατάσταση, έχει υποστεί σοβαρές ρογμές το αυταρχικό στερέωμα του αραβικού κόσμου. Θέλω τώρα να σταθώ σε ορισμένε συγκεκριμένες χώρες στον Περσικό κόλπο και να αναφερθώ επίσης και στο ευρύτερο θέμα του αραβικού κόσμου. Στην περίπτωση της Λιβύης, δυστυχώς, αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση τελμάτωσης, μια κατάσταση όπου δεν υπάρχει πλεονέκτημα ούτε της μιας είτε της άλλης πλευράς και ολισθαίνει η Λιβύη σε μια παρατεταμένη διαμάχη και σύγκρουση και όχι σε μια μετάβαση σε ένα νέο μέλλον. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εύκολος τρόπος για να μπορέσει κανείς να βγει από αυτό το αδιέξοδο στη Λιβύη. Οι περισσότεροι από εμά έχουμε υποτιμήσει όχι μόνο την αντοχή του Καντάφη και της φατρίας τους και την αποφασιστικότητα του συνταγματάρχη Καντάφη να αγωνιστεί ως το τέλος. Έχουμε επίσης υποτιμήσει μέσα στη Λιβύη το ότι η Λιβύη είναι μια πολύ πιο διηρημένη κοινωνία από ό,τι περισσότερο από εμά ελπίζαμε να είναι. Και επειδή περισσότερο από εμά θεωρούμε ότι είναι ένας κακός και βίαιος άνθρωπος ο κύριος Καντάφη, κάπου βολευτήκαμε όλοι σε μια συλλογική μορφή σκέψης που μας έκανε να πιστεύουμε ότι σε λίγες μέρες, σε λίγες βδομάδες θα ξεπεραστεί. Αλλά δεν έχουμε λάβει υπόψη τη βαθιά, το βαθύ διχασμό που υπάρχει στη Λιβύη. σημαίνει αυτό ότι ο Καντάφη έχει μια ευρεία υποστήριξη, αλλά ο συνταγματάρχης Καντάφη έχει μια περιορισμένη αλλά πολύ ισχυρή βάση υποστήριξης. Αυτή η ισχυρή βάση υποστήριξης η οποία απαρτίζεται από ορισμένε φυλές από επαναστατικές επιτροπές, γιατί μιλάμε για ένα καθεστώς το οποίο είναι στην εξουσία εδώ και 41 χρόνια και ουσιαστικά έχει προσετεριστεί ένα μεγάλο αριθμό ατόμων και έχει ισχυρές δυνάμεις, ε, ειδικές δυνάμεις το κράτος και έχει τους γιους του που είναι επικεφαλής αυτών των ειδικών δυνάμεων και έχει μαζί του τους ηγέτες πολλών φυλών. Έχουμε λοιπόν μια περιορισμένη αλλά ισχυρή βάση υποστήριξης ε, του Καντάφη, η οποία αντιμετωπίζει και μία ανίκανη αντιπολίτευση. Δυστυχώ είναι πολύ πιο ανίκανη η αντιπολίτευση από ό,τι την περιμέναμε να είναι. Δεν πρέπει να είμαστε τόσο σκληροί ίσω μαζί του, γιατί αυτή η αντιπολίτευση έχει μονάχα έξι εβδομάδε ζωή. Αλλά δεν μπόρεσε αυτή η αντιπολίτευση στον Καντάφη να χρησιμοποιήσει τις, ε, τα πλήγματα που καταφέρθηκαν κατά του Καντάφη τις τελευταίες εβδομάδες από την συμμαχία εναντίον του. Αυτό καταδεικνύει και το βάθος της κρίσης στην Λιβύη. Αν η αντιπολίτευση, αν οι αντίμαχοι του Καντάφη δεν μπόρεσαν να υποφεληθούν από τα κέρδη που πέτυχαν τι προηγούμενε εβδομάδε, αμφιβάλλω πάρα πολύ αν υπάρχει κάποια διέξοδο από την τονική κατάσταση στη Λιβύη. Ο φόβο μου είναι ότι όσο σοβεί αυτή η κρίση στη Λιβύη, όσο περισσότερο χρόνο κρατά αυτή η κρίση, τόσο περισσότερο θα βυθιστεί η Λιβύη, όχι μόνο σε μια παρατεταμένη σύγκριση, σύγκρουση, αλλά κυρίως σε ένα παρατεταμένο ε, εμφύλιο πόλεμο. Αυτό είναι το χειρότερο λοιπόν σενάριο, ένα σενάριο που θα οδηγήσει στην κατάρρευση της Λιβύης με έναν τρόπο αντίστοιχο του Αφγανιστάν και της Σομαλίας. Μου φαίνεται λοιπόν ότι η κατάσταση στη Λιβύη είναι πάρα πολύ πολύπλοκη, πολύ εύθραυστη και ευαίσθητη και δεν πρόκειται στο άμεσο μέλλον να αποχωρήσει ο συνταγματάρχης Καντάφη. Από όλα αυτά που ξέρουμε για το Καντάφη, είναι φανερό ότι θα παραμείνει και θα πολεμήσει μέχρι τον τελευταίο άντρα, μέχρι την τελευταία ε, σφαίρα και θα πει στο τέλος από θανέτου η ψυχή μετά των άλλων φίλων. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να γεμίσουμε, να δώσουμε κάποιο περιεχόμενο στην ε, πολιτική κατάσταση στη Λιβύη, παρά το γεγονό ότι όλοι θέλουμε να φύγει ο Καντάφη, βλέπουμε ότι η Αφρικανική Ένωση κάνει μια προσπάθεια διαμεσολάβησης. Θα έπρεπε η Ιταλία, πιστεύω, και η Γερμανία και τα Αραβικά κράτη και η Αφρικανική Ένωση να κάνουν μια προσπάθεια να φέρουν σε επαφή και αυτούς που παραμένουν πιστοί στον Καντάφη, αυτοί που είπα ότι είναι περιορισμένοι αλλά ισχυροί οπαδοί του Καντάφη. Γιατί ακόμα και αν φύγει ο Καντάφη ο ίδιος, η επαύριο θα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ επικίνδυνη. Γι' αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι υπέρμαχοι του Καντάφη και να έρθουμε σε επαφή μαζί τους για το καλό της Λιβύης, για το καλό των Λίβιων, για το καλό της σταθερότητας σε αυτό το τμήμα του κόσμου. Και τώρα να έρθω σε ένα άλλο σημείο για την Ιεμένη και συγγνώμη αν, ε, αν απλοποιώ πάρα πολύ τα πράγματα. Είναι πάρα, πάρα πολύ δύσκολη η επιλογή. Ή ο Αλσαλέχ θα αποχωρήσει ή αλλιώς η Εμένη θα βρεθεί και αυτή σε μια αντίστοιχη κατάσταση με αυτή που βλέπουμε στη Λιβύη. Θέλω να προχωρήσω όμως και περισσότερο. Θέλω να προχωρήσω για να πω ότι ένας εμφύλιος πόλεμος στην Ιεμένη θα είναι ακόμα πιο επικίνδυνος από αυτό που βλέπουμε σήμερα στη Λιβύη. Η Ιεμένη είναι μια πολύ πιο επικίνδυνη κατάσταση, μια πολύ πιο εύθραυστη χώρα όχι μονάχα γιατί έχετε πολλές διαιρέσεις σε φιλετική ε, βάση. Ξέρετε ότι υπήρχε στο παρελθόν μια, ένα αποσχιστικό κίνημα στο Νότο, είχατε μια εξέγερση στο Βορρά, μια ισχυρή βάση της στην κεντρική Ιεμένη. Από όλα αυτά τα οποία γνωρίζουμε λοιπόν για την Ιεμένη, η βάση της Αλκάιντα στην Ιεμένη πολύ πιο ισχυρή από την κεντρική βάση της Αλ-Κάιντα στις ε, περιοχές που έχουν το φιλετικό δίκαιο στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Από ό,τι ξέρουμε λοιπόν για τον πρόεδρο Αλ Σαλέχ, φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμος να αποχωρήσει και χαίρομαι για το γεγονός ότι ακόμα και η αμερικανική εξωτερική πολιτική έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι πρέπει παρόλα αυτά να φύγει ο πρόεδρος Αλ Σαλέχ, γιατί η ίδια η παρουσία του δημιουργεί το σπινθήρα ο οποίο θα οδηγήσει σε μία μίζωνα ανάφλεξη στην ίδια την Ιεμένη. Και ο λόγος για τον οποίο η κατάσταση εκεί έχει κλιμακωθεί σε ένα τόσο επικίνδυνο επίπεδο, όπως ξέρετε είναι χωρισμένο στα δύο στρατός, ιδίως ε, μεταξύ των ειδικών δυνάμεων τον οποίο ηγείται ο γιος και οι συγγενείς του Πρόεδρου Αλσαλέχ και που αρρωγείται από ορισμένες ειδικέ δυνάμεις ε, από τη δική του φίλη και υπάρχει αυτή η σύγκρουση μεταξύ των ειδικών δυνάμεων του Αλσαλέχ και αυτών που έχουμε αποχωριστεί από το στρατό. Και αυτό σας δείχνει ότι η κατάσταση ασφάλειας γίνεται ακόμα πιο επισφαλής τα τελευταία τις τελευταίες εβδομάδες. Έχουν γίνει σημαντικές επιθέσεις από την Αλκάιντα σε εργοστάσια παραγωγής πυραμαχικών και είναι σαν να περιμένει η Αλκάιντα στην Ιεμένη για την κατάλληλη στιγμή να δράσει. Αυτό βέβαια δεν είναι ένα πρωτότυπο ε, επιχείρημα. Ξέρουμε ότι η Αλκάιντα τρέφεται με την κοινωνική αστάθεια. Αν υπάρξει λοιπόν εμφύλιο στην Ιεμένη, ή μάλλον πολλαπλή εμφύλη, μπορείτε να καταλάβετε τι συνέπειε, όχι μόνο για την Ιεμένη. Η Ιεμένη έχει ένα τεράστιο, μια τεράστια συνοριακή γραμμή με τη Σαουδική Αραβία. Όλες οι συνολικές λοιπόν από όλε τι συνολικέ απειλέ ασφάλεια προ τη Σαουδική Αραβία, πιστεύω ότι η μεγαλύτερη είναι αυτή η οποία μπορεί να προέρχεται από την Ιεμένη. Κίνδυνο, όχι μονάχα για το βασίλειο της Σαουδική Αραβίας, αλλά και για όλη αυτή την περιοχή, γιατί υπάρχει το δυναμικό, η δυνατότητα να εκμεταλλευτεί κάποιο τις διαφωνίε και διαμάχες μεταξύ των φινών. Θυμόσαστε ότι η, η Εμένη ήταν, χάρη στον πρόεδρο Σαλέχ, μία από τις πιο, από τις λιγότερο σεχταριστικές ήταν λιγότερο, μια από τι λιγότερε εκταριστικέ κοινωνίε στον κόσμο, αλλά επειδή εκμεταλλεύτηκε τι διαιρέσει Ιητών και Σουνιτών, ο Αλσαλέχ τώρα είναι μια από τι πιο εκταριστικέ χώρε στον κόσμο. Η κατάσταση λοιπόν στην Ιεμένη θα μπορούσε να κλιμακωθεί προ το χειρότερο. Χρειάζεται απλώ ένα πινθήρα, όπω είπα, και υπάρχει αυτή η κατάσταση όπου έχουμε μια υποβόσκουσα σύγκρουση σε όλο το έδαφο τη Ιεμένη. Θα πρέπει να δούμε αν ο πρόεδρο Αλσαλεχ θα ακούσει τι φωνέ της λογικής και της οφροσύνη μέσα στη χώρα του, στην ευρύτερη περιοχή και στη διεθνή κοινότητα και θα δεχτεί μια λύση βάσει της οποίας θα υπάρξει μια ειρηνική μετάβαση για την εξουσία στην Ιεμένη. Έρχομαι στο Μπαχρέιν. Χαίρομαι για τη δήλωση του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σήμερα. Είναι μια αποφασιστική δήλωση, πιστεύω, και μια δήλωση η οποία είναι εύγλωτη για την κατάσταση του Μπαχρέιν. Παρά το γεγονό ότι θα έλεγα ότι η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και οι σκληροπυρονικοί στον Μπαχρέιν έχουν κερδίσει τον πρώτο γύρο, η κατάσταση δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει. Θα υπάρξει δεύτερος γύρος, θα υπάρξει και τρίτος γύρος και αν δεν αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση και όταν λέω αντιμετωπιστεί αν δεν υπάρξει πλήρης διαδικασία διαλόγου μεταξύ της βασιλικής οικογένειας και της αντιπολίτευσης, δεν πρόκειται να περατωθεί αυτή η κρίση στο Μπαχρέιν. Αυτό το οποίο αποτελεί ηρωνία είναι ότι αυτή τη στιγμή η αντιπολίτευση στο Μπαχρέιν δεν ζητούν τον ουρανό μετάστρα. Ζητούν απλώς να υπάρξει μια δυνατότητα να συμμετάσχουν στον πολιτικό και κοινωνικό χώρο, να έχουν τη δυνατότητα να γίνουν αποδεκτοί, να έχουν τη δυνατότητα να έχουν θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα και στις δυνάμεις ασφαλείας, να υπάρχουν συνταγματικές αλλαγές οι οποίες θα φέρουν τον Μπαχρέν σε μια, σε μια κατάσταση πιο διαφανούς κοινωνίας και να, μιας κοινωνίας με πιο διάφανες μορφές εξουσίας. Δυστυχώς όμως αυτά δεν γίνονται τώρα γιατί οι σκληροπυρηνικοί στο Μπαχρέν έχουν κερδίσει το πάνω ε, με τη βασιλική οικογένεια και ο φόβος μου, ο λόγος που και εγώ ανησυχώ για τον Μπαχρέν όπως και πολλοί άλλοι, ο φόβος μου είναι ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη ριζοσπαστικοποίηση στη χώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή βράζει η χύτρα μετά από τη βία καταστολή που έγινε της αντιπολίτευσης στον Μπαχρέν. Φοβόμαστε επίσης ότι η όξυνση των ε, ε, διαμαχών στη, στο Μπαχρέν μπορεί να γίνει ακόμα μεγαλύτερη. Βλέπουμε όλο και περισσότερο πόσο σεχταριστική γραμμή κράτησε η αντιπολίτευση που στην αρχή είχε προσπαθήσει να παρουσιάσει μια ορθολογική εικόνα του εαυτού της. Υπάρχει κίνδυνος ότι λοιπόν θα μπορούν να γίνουν χειρότερα τα πράγματα στον Παχρέν. Υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος ότι το Ιράν μπορεί να το βρει πολύ ευκολότερο να αναμειχθεί στην κρίση στον Παχρέν με την τεράστια καταστολή που ασκείται από τη βασιλική οικογένεια στον Μπαχρέν. Πιστεύω λοιπόν ότι η κρίση στον Μπαχρέν έχει ένα κρίσιμο ρόλο. Εφόσον βρισκόμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη Δύση να δείξει μια συνεκτική στάση. Γι' αυτό η δήλωση του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δεν μπορούμε από τη μία πλευρά να λέμε, να πουλάμε εξοπλισμού στη Λιβύη και να ε, μην είμαστε συγχρόνως σαφής για τη θέση που έχουμε σε σχέση με την οποιαδήποτε χώρα. Είναι μια κρίσιμη στιγμή για τη Δύση, είναι μια στιγμή που πρέπει να την αδράξουμε και να δείξουμε ότι η Δύση ενδιαφέρεται για τη δημοκρατία, ότι η Δύση είναι στην προοδευτική πλευρά της ιστορίας και αυτά που γίνονται στον Παχρέν έχουν σημασία όχι μόνο για τους πολίτες του Παχρέν αλλά για τη σύνολη διεθνή κοινότητα. Και πιστεύω και πάλι, όπως ξέρετε, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια κρίση μεταξύ Σαουδική Αραβία και Ηνωμένων Πολιτειών στους τελευταίους τρει μήνες, όχι μόνο λόγω του Μπαχρέιν <clears throat> και όχι μόνο λόγω τη κατάσταση στην Αίγυπτο και την Τινησία. Η Σαουδική Αραβία πιστεύει ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν βοηθήσει τους συμμάχους τους, έχουν αφήσει τους συμμάχους τους αποήθου, ακόμα και του έχουν μαχαιρώσει στην πλάτη και οι Ηνωμένε Πολιτείε πιστεύουν δεν υπάρχει καμία δυνατότητα λύση χωρί μείζονε μεταρρυθμίσει σε αυτή την περιοχή. Στην περίπτωση όμω του Μπαχρέιν, οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν έχουν υψώσει τη φωνή του όσο θα έπρεπε να το είχαν πράξει και οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν επιτρέψει στη Σαουδική Αραβία να κερδίσει τον πρώτο γύρο αντιπαράθεση στο Μπαχρέν, γιατί σύμφωνα με του υπολογισμού τη κυβέρνηση Ομπάμα, η σχέση Πολιτειών και Σαουδικής Αραβίας παίζει πιο σημαντικό χαρακτήρα, πιο αξονικό χαρακτήρα έχει από ότι οι δημοκρατικές προσδοκίε τη αντιπολίτευσης στο Μπαχρέν και γενικά στον Περσικό κόλπο. Και θέλω εδώ να <clears throat> αναφερθώ, εφόσον μιλάμε για τον Περσικό κόλπο, ότι παρά το γεγονός εγώ δεν πιστεύω ότι η Σαουδική Αραβία είναι τόσο τρωτή όσο τα κράτη της Βόρειας Αφρικής ή όπως το ίδιο το Μπαχρέιν ή η Λιβύη ή η Εμένη. Η Σαουδική Αραβία δεν είναι άμομη από τις δυνατότητες να μολυνθεί μέσα σε εισαγωγικά από το δημοκρατικό ιό της περιοχής. Δεν είναι απόλυτα προστατευμένη η Σαουδική Αραβία παρά το γεγονός ότι δεν είναι τόσο τρωτή όσο άλλες χώρες. και νομίζω πρέπει να σκεφτούμε για το βασίλειο της Σαουδικής Αραβίας για πολλούς λόγους. Υπάρχουν οι προσδοκίες των νεαρών Σαουδαράβων που δεν διαφέρουν πάρα πολύ από τις διεκδικήσεις των νέων που βρίσκονται σε άλλες χώρες της ε, περιοχής. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι νέοι στη Σαουδική Αραβία, μερικοί από τους οποίους είναι φοιτητέ μου, έχω διδάξει στο Κολούμπια, στις Ηνωμένες τώρα είμαι στο London School of Economics, δεν βλέπω λοιπόν να υπάρχουν διαφορές ουσιαστικές μεταξύ των Σαουδαράβων νέων, των Αιγυπτίων, των Ιεμενών, αυτών που προέρχονται από την Ιεμένη ή την Θέλουν περισσότερη δημοκρατία, πιο διάφανη κοινωνία, ενοχλούνται πάρα πολύ από την ευρύτητα και την έκταση της διαφθοράς, όπως και οι άλλοι νέοι σε χώρες της, ε, της, ε, του αραβικού κόσμου. Τα νέα μέσα ε, επικοινωνία τα κοινωνικά δίκτυα και όλα αυτά έχουν διαβρώσει <clears throat> και τον έλεγχο της κυβέρνησης. Γιατί πια ο πληθυσμό Σαουδικής Σαουδική έχει πρόσβαση σε πολλαπλέ μορφέ πληροφόρηση και αυτό έχει αλλάξει τι ισορροπίε μέσα στο, στη Σαουδική Αραβία. Όπω και στον Παχρέν. Υπάρχει μια μεγάλη κοινότητα στην Σαουδική Αραβία που θεωρεί ότι είναι αντικείμενο διάκρισης. Μιλάμε για ένα περίπου 20% του πληθυσμού της Σαουδικής Αραβίας. Γι' αυτό η ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας παρενέβη στον Παχρέν γιατί ο φόβος της ήταν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στον Παχρέν θα μπορούσε να επηρεάσει και τις ε, συνθήκες στο, στις ανατολικές επαρχίες της Σαουδικής Αραβίας θα επιχειρηματολογούσα εδώ, ίσως κάνω λάθος, ότι η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας δεν έχει κατανοήσει ακόμα τη σοβαρότητα της κρίσης. Η ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας είναι σαν τη στουρδοκάμιλο, θάβει το κεφάλι της στην άμμο, ενώ η αμερικανική κυβέρνηση ξέρει πόσο σοβαρή είναι αυτή η κρίση, είπε η Αμερικανική κυβέρνηση εντάξει δεν πειράζει και άφησε τους Σαουδάραβες να κάνουν αυτό το οποίο πιστεύουν γιατί είναι πάρα πολύ στενή η σχέση της Σαουδικής Αραβίας με την κυβέρνηση Ομπάμα και η Ομπάμα και οι δικοί του θεώρησαν ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή να έρθει σε σύγκρουση με την Σαουδική Αραβία όταν υπάρχει μια εξέγερση στη συνολική περιοχή. Και πάλι δεν πρόκειται μοναχά για τον Μπαχρέιν αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε και το δεύτερο και τον τρίτο γύρο στο Μπαχρέιν. Δεν θα πρέπει να πάρουμε για δεδομένη την εσωτερική κατάσταση στη Σαουδική Αραβία, γιατί και πάλι ο ιός της δημοκρατίας αλλάζει μορφή και πηγαίνει από χώρα σε χώρα. Πολλοί από μας πιστεύανε ότι αυτό το πράγμα θα μπορούσε να φτάσει μέχρι και τη Συρία. Εγώ ποτέ μου δεν είχα φανταστεί ότι δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες Σύριοι θα τολμούσαν να αψηφίσουν τις κυβερνητικές δυνάμεις στους δρόμους. Δείχνει λοιπόν πραγματικά ότι κάτι έχει συνεπάρει τον κόσμο σε αυτή την περιοχή, ότι έχει ξεπεραστεί ο παραγόν φόβος. Κάτι σημαντικό έχει γίνει λοιπόν στην περιοχή αυτή. Και μου λένε ότι έχει τελειώσει ο χρόνος μου, θα κλείσω εδώ και απλώς θέλω να πω μόνο για ένα λεπτό να πω δύο, δύο πράγματα για το τι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορούν να κάνουν. Πιστεύω ότι αν υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα που θέλω να τονίσω, είναι ότι από θεσμική άποψη η Μέση Ανατολή είναι μια έρημος. Ιδίω ο αραβικός κόσμος είναι μια έρημος σε ό,τι αφορά τους θεσμούς. Από όλους τους φορείς λοιπόν που υπάρχουν αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν τη μεγαλύτερη δυνατότητα να παίξουν ένα κρίσιμο ρόλο για να βοηθήσουν τη διαδικασία οικοδόμησης θεσμών στην περιοχή αυτού του κόσμου με τον να έρθουν σε επαφή με τις αναδυόμενες δυνάμεις σε πολλαπλά επίπεδα δίνοντας υποτροφίες, χορηγίες, σεμινάρια συμφιλίωσης, ανταλλαγές, ε, υποστήριξη μέσων ενημέρωσης να βοηθήσουν τις νέες δυνάμεις που αναδύονται στην περιοχή αυτή να οργανωθούν καλύτερα και να δημιουργήσουν ένα αντίπαλο δέος στις κυρίαρχες δυνάμεις που είναι οι οργανωμένες αυταρχικές οι αυταρχικές δυνάμεις και επίσης τους Ισλαμιστές, γιατί οι Ισλαμιστές στην Ιεμένη, στη Λιβύη, στην Αίγυπτο είναι αυτή τη στιγμή οι πιο ισχυροί και οι πιο οργανωμένοι αντίπαλοι των καθεστώτων. Και δεν σας λέω ότι πρέπει να ανησυχήσουμε πάντα για όλες τις Ισλαμικές δυνάμεις, αλλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει τις δυνάμεις του κέντρου, τις κοσμικές δυνάμεις να ενισχύσουν τον εαυτό τους και να πάρουν τη δυνατότητα να έχουν τους κατάλληλους θεσμούς στις χώρες τους. Θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστούμε. Ε, δεν είναι εύκολο να καλύψει κανείς μια τέτοια περίπλοκη κατάσταση, αλλά τα καταφέρατε. Ευχαριστούμε για την ε, συνεκτικότητα και την ε, ε, ουσιαστικότητα των αυτών που είπατε. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Νίμπλερ. έτσι είχαμε συμφωνήσει να λάβετε το λόγο και μπορείτε να αντλήσετε και τα συμπεράσματα στο τέλος. Αν θέλετε να λάβετε τώρα το λόγο, επίσης μπορείτε. Σας ευχαριστώ μου δίνετε την ευκαιρία να λάβω και τώρα το λόγο και κύριε Γκέργες. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας μεταφέρατε τις απόψεις σας για όλη αυτή την περιοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω λοιπόν για τον διαφοροποιημένο τρόπο με το οποίο παρουσιάσατε την κατάσταση και στη Λιβύη και στην Ιεμένη και στον Παχρέν και στη Σαουδική Αραβία. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίζουμε αυτά τα γεγονότα όχι ισοπεδωμένα με τον ίδιο τρόπο, αλλά με διαφοροποιημένα ανάλογα με την κάθε χώρα και την κάθε περιοχή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη συζήτηση τη Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχουμε μια διαφοροποιημένη άποψη για τα θέματα αυτά. Κάποιε προκαταρκτικέ παρατηρήσει. Από τη δική μου πλευρά, λέτε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να δείξουν μια συνεκτικότητα και συνέπεια στην τοποθέτησή του κατά του έναντι του αραβικού κόσμου και είμαι πάντα είμαι απόλυτα σύμφωνοι μαζί σα. Εμεί ω Κοινοβούλιο θεωρήσαμε ότι πάντα πρέπει να δώσουμε έμφαση στη δημοκρατία, στο κράτο δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, να αγωνιστούμε για τα θέματα αυτά και δεν έχει αλλάξει η στάση μα αυτή. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και για αυτή τη δήλωση που έκανε ο πρόεδρο μα σήμερα. Εγώ μίλησα με τη συνάδελφο Χάιντι Χάουταλα, η οποία είναι η πρόεδρο τη Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και κάναμε και <clears throat> μια κοινή δήλωση σε σχέση με τις επιθέσεις στο Μπαχρέν, τις οποίες καταδικάζουμε στεναρά και δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να κατηγορήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι δεν ξέρει σε ποια πλευρά βρίσκεται. Στην τελευταία μας συνάντηση εδώ πέρα είχαμε και ένα εκπρόσωπο της Κομισιόν ο οποίος όπως και, εσάς, και εσείς παρουσίασε μια κατάσταση της, ε, μια, μια έκθεση της ε, επιτόπιας κατάστασης. Υπήρξαν πολλές κριτικές απόψεις από τους συναδέλφους γιατί θέλαμε τον κύριο Κούπερ από τον, πρόεδρο από τον εκπρόσωπο της Κομισιόν να ε, απαντήσει στα <clears throat> ερωτήματά μας και στην περίπτωση του Μπαχρέν είπε απλώς ότι ήταν μια κατάσταση δυνάμει εμφυλίου πολέμου. Δεν είχε λοιπόν παρουσιάσει τα πράγματα με, τόση, με τόσο λεπτολόγο τρόπο όπως και εσείς. Όταν λοιπόν έχουμε προβλήματα με την ε, σταθερότητα της αντίληψης που έχουμε για τα ζητήματα αυτά, αυτό είναι περισσότερο ένα διαθεσμικό πρόβλημα. Το Κοινοβούλιο έχει πάντα μια σταθερή στάση για τα πρόβληματα αυτά. Και μια τελευταία παρατήρηση ως πρόεδρος της αντιπροσωπείας για την ε, Αραβική Χερσόνησο. Ήμασταν πρόσφατα στην περιοχή αυτή, πήγαμε στη Μανάμα, περάσαμε και κάποιο χρονικό διάστημα στο Κουβέιτ και είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε και το Κοινοβούλιο του Κουβέιτ και ήρθε, προσκαλέστηκε και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Κουβέιτ εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και νομίζω ότι αυτά τα οποία προτείνατε εσείς για τις επαφές με την κοινωνία των πολιτών και την υποστήριξή της είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πρέπει να δημιουργήσουμε υποστηρικτικές δομές οι οποίες θα μπορέσουν να ανοίξουν το δρόμο για τη δημοκρατία στις περιοχές αυτές. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ θετικέ οι επαφές μας με το Κουβέιτ που έχει ένα ιδιαίτερα ζωντανό και έντονο κοινοβουλευτικό βίο μπορέσαμε να λάβουμε μέρος σε μια συζήτηση εκεί. Είδαμε ότι υπάρχουν πολλές γυναίκες μεταξύ των εκλεγμένων εκπροσώπων στο Κουβέιτ. Αυτό είναι ήδη μια πρόοδο. Υπάρχει μια κίνηση σε αυτή την περιοχή ώστε να κινηθούν οι χώρες αυτές προς τη σωστή κατεύθυνση και αυτό πρέπει να το υποστηρίξουμε. Τελευταία μου ερώτηση σε εσά. Σκεφτόμενοι πάλι την Ευρωπαϊκή Ένωση, σκεφτόμενοι πάντα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μας είπατε τι είναι αυτό που θεωρείτε ότι είναι σημαντικό για σας. Θα ήθελα να ξέρω το εξή, Το Συμβούλιο Συνεργασίας του Περσικού Κόλπου, κατά την άποψή σα τι ρόλο θα έπρεπε να παίξει. Γιατί δεν είναι <clears throat> οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν μια συνεργασία για την εξασφάλιση της ασφαλείας και αναφερθήκατε ιδιαίτερα στο θέμα της Σαουδικής Αραβίας που έστειλε μαζί με τα άλλα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας στρατιωτικά αγίματα στον Παχρέν Αλλά ποια θα μπορούσε να είναι η συμβολή αυτής της κοινότητος για να εξασφαλίσει περισσότερη σταθερότητα στην περιοχή αυτή και μια τακτικού χαρακτήρα και μια συντεταγμένη μετα... μεταρρύθμιση εκεί. Λόγω του χρόνου των ατόμων που ζήτησαν το λόγο και λόγω των περιορισμών που έχουμε, οφείλω να περιορίσω σε τρία λεπτά τον λόγο που θα έχετε στη διάθεσή σας. Ο κύριος Ενσκίνς. Συγγνώμη, δεν άκουσα το ότι είπατε τρία λεπτά, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ε, συγχαρώ για όλα όσα είπατε. Υπάρχουν τόσα θέματα, τόσες ερωτήσεις που μπορώ να θέσω που δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Καταρχήν δεν ξέρουμε ποιο θα είναι το μέγεθος το οποίο θα αποφασίσουμε να κρατήσουμε. Θέλουμε να επιλέξουμε καταρχήν ή την σταθερότητα ή τη δημοκρατία. Γιατί αν ε, στο παρελθόν είχαμε τη σταθερότητα ως γνώμονα στην Μέση Ανατολή, τώρα δεν ξέρουμε εάν μέσω ημών να αναπτυχθεί αυτός ο τομέας γιατί αυτόν θέλουμε πιο πολύ από να ε, φροντίσουμε. Ε, επίσης ε, μου φαίνεται πάρα πολύ σαφές σε αυτήν την ε, αφύπνιση της Μέσης Ανατολής το ότι η Κάιτα είναι κάτω από, την, από το Χαμάς. Υπάρχουν παίκτες πολύ σημαντικοί και οι οποίοι καθοδηγούν, είναι ηγέτες ας πούμε της Επανάστασης. Άλλοι ε, εκτός από αυτά τα Ισλαμιστικά σώματα, τα εξτρεμιστικά. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό, για το αν υπάρχουν και ποιοι είναι και επίσης το θέμα της ε, θεσμικής υποστήριξης. Το θέμα είναι ότι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ένας παρατηρητής και όχι ένας παίκτης μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να αναπτύξουμε μια θεσμική στήριξη με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να μην δίνουμε απλώς χρήματα του φορολογουμένου για να τους στηρίξουμε, περιμένοντας την απάντησή σας.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 ε, κάτι που έχει σχέση με τις ερωτήσεις του... Μάλλον συμμερίζομαι και εγώ τις ερωτήσεις του κυρίου Άτκινς. Ε, ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τι συνεισφορά μπορεί να προσφέρει, όπως έχει κάνει σε άλλες χώρες. Ε, βεβαίως αυτό καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι που είναι βραχυπρόθεσμο. Είναι κάτι που θα διαρκέσει πολύ καιρό. Ε, Πώς θα γίνει να έχουμε ένα βιώσιμο κράτος το οποίο, θα μπορέσουμε μετά να, το οποίο θα μπορέσει μετά να πάρει την πορεία του. Όχι, Όσο αφορά την ε, διαμεσολάβηση της Αφρικανικής Ένωσης, αν θα δείτε ότι δεν ε, είναι καθόλου πιστική. Δεν ξέρουμε αν κάτι μπορεί να προκύψει από αυτό. Έχουν υπάρξει λοιπόν υποστηρίξεις με σημαντικά κονδύλια των περιοχών αυτών και βλέπουμε ότι η στάση του Ζούμα ε, του από την Νότια Αφρική που λέει δεν πάω στη Βενγάζη γιατί έχω καλύτερα πράγματα να κάνω στη ζωή μου Έχουμε πάρει λοιπόν... Έχουμε πάρει λοιπόν και μία πρόγευση από αυτά τα οποία μπορούν να προκύψουν από την ε, αντιμετώπιση λοιπόν της ε, Αφρικανικής Ένωσης. Τι έχετε να πείτε σε σχέση με αυτό. Ευχαριστώ κύριε. Ο κύριος Φόξ για τρία λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ ε, για αυτήν την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Θα ήθελα να σχολιάσετε για τη σημασία του γεγονότος ότι η Αραβική Λιώνα ψήφισε ε, υπέρ μιας ζώνης e uh, μια ζώνης μη υπέρπτυσης ε, υπάρχει μια απόφαση ανάληψη στρατιωτικών επιχειρήσεων και η ηγετική θέση σε αυτή την απόφαση ήταν ε, της Γαλλίας και η Γερμανία δίσταζε πάρα πολύ παρά ε, το γεγονός ότι η Αραβική Λίγκα είχε ζητήσει δράση και δεν ενισχύεται έτσι το γεγονός ότι η κοινή ε, πολιτική, ευρωπαϊκή, εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας είναι κάτι που παραμένει ε, στα κράτη-μέλη ε, γενικά και αυτά τα γεγονότα που τα τελευταία το υπογραμμίζουν αυτό το φαινόμενο. Τι λέει το υπόλοιπο του κόσμου και ειδικά ε, ο αραβικός κόσμος σε σχέση με την ΕΕ. Αν αυτά που είδαν τις τελευταίες έξι, εβδομάδες, τις τελευταίες έξι εβδομάδες υπάρχει ένα πρόβλημα εάν δεν είναι δυνατόν να δράσουμε ενοποιημένα ακόμα και όταν οι αραβικοί τότε ε, νομίζω ότι έχουμε ε, εντελώς διαμοιράσει ε, το, την ε, ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας. Ε, τι μπορεί να κάνει λοιπόν θετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην διαλυθεί αυτό το κράτος. Είμαστε απλοί παρατηρητές και τίποτε άλλο δηλαδή. ευχαριστώ πολύ κύριε Φόξ. Ο κύριος Γιατεμάκη, η κυρία Γιατεμάκη για τρία λεπτά. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για το, τον αποκλεισμό των όπλων. Ε, το, σχετικά με τον συνταγματάρχη Καβα, Καντάφη. Συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι είναι πάρα πολύ ισχυρός γιατί έχει πάρα πολύ καλές ε, θέσεις και ισχυρή υποστήριξη γιατί του πούλησαν ε, όπλα στον Καντάφη οι ευρωπαϊκές δυνάμεις για πάρα πολλά χρόνια του πουλούσαν όπλα και ακόμη και φέτος οι μεγαλύτερες εξαγωγές ε, έγιναν με τους εμπειρογνώμονες οι οποίες έδιναν συμβουλές στα σώματα στις ομάδες ασφαλείας. Θα πρέπει τώρα λοιπόν να πάψουν να χρησιμοποιούν τα όπλα τους. Ναι, αλλά ε, αφού γίνεται, γίνονται πωλήσει όπλων. Νομίζω λοιπόν ότι το πιο σημαντικό θέμα για την ευρωπαϊκή πλευρά θα ήταν επιτέλους να σταματήσει να πουλάει όπλα σε αυτές τις αραβικές χώρες. Τέλος πάντων μπορείτε να μας πείτε με δυο λόγια τι πιστεύετε, τι φρονείτε για αυτό το θέμα της πώληση των όπλων. Ε, και Πέρα από αυτό θα ήθελα να ακούσω κάτι παραπάνω για την ιστορία της Λιβύης. Δεν νομίζω αν είναι αλήθεια, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, αλλά κατάλαβα ότι κατά την περίοδο της ε, απικιοκρατίας υπήρχαν ε, ε, πολλά τμήματα, πολλά μέρη, δεν, δεν ήταν ενοποιημένη η κατάσταση και το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει μια κληρονομιά αυτή τη κατάσταση και ότι υπάρχουν μεγάλες ομάδες που είναι υπέρ του Καντάφη και μεγάλες ομάδες κατά του Καντάφη. Και αυτό είναι κομμάτι της ιστορίας της Λιβύης νομίζω. Ε, ευχαριστώ πολύ για την ανακοίνωσή σας. Ευχαριστώ κυρία Γιατεμάκη. Ο, ο λόγος του κύριο Αρλάκη. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια καθηγητά για τη σαφήνεια και το βάθος της ανάλυσης. Έχω 42 ερωτήσεις. Θα περιοριστώ στις πρώτες πέντε. Για την κατάσταση στις χώρες του κόλπου και της Μέσης Ανατολής. Πρώτον, Πώς πιστεύετε θα εξολιχθεί αυτό το δεύτερο κύμα εκδημοκρατισμού, το κύμα που τώρα υψώνεται στα Εμμυράτα, τη Σαουδική Αραβία και τις χώρες που έχουν απομείνει. Βλέπετε να υπάρξει κάποια εξέλιξη προς συνταγματική μοναρχία, προς συνταγματικές μοναρχίες. Βλέπετε μια μη βίαιη σύγκρουση μια μη βίαιη αντιπαράθεση. Δεύτερη ερώτηση για τους εξοπλισμούς ε, στο, στις χώρες του κόλπου. Ε, γνωρίζουμε ότι είναι η πιο οπλισμένη περιοχή στον κόσμο. Η Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα οι χώρες συνεργασίας του κόλπου, απορροφούν το 50% των παγκόσμιων ε, προϋπολογισμών για τους εξοπλισμούς. Η ιδέα ενός εμπάργου πώλησης όπλων. Ε, θέλουμε να μειωθεί ο προϋπολογισμός ε, των χωρών αυτών ε, για τους εξοπλισμούς. Πιστεύετε ότι αυτό θα, θα επηρεάσει θετικά, θα, πιστεύετε ότι θα επηρεάσουμε θετικά την κατάσταση με ένα εμπάρκο. Οι πολιτές ε, όπλων, ιδέως από τις Ηνωμένε Πολιτείε και τους Βρετανούς, είναι οι πιο σημαντικοί πολιτές όπλων, προμηθευτές όπλων στην περιοχή εμπάργκο όπλων ε, ίσως δικαιολογείται στην περίπτωση της Ιρανικής απειλής. Η Ιρανική απειλή πιστεύω ότι είναι το μείζον στοιχείο που δικαιολογεί το τεράστιο ποσό χρημάτων που πηγαίνουν στους εξοπλισμούς. Εσείς πώς αξιολογείτε την Ιρανική απειλή. Θεωρείτε ότι δικαιολογεί τις στρατιωτικές δαπάνες. Η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία. Φυσικά υπάρχει το μεγάλο ζήτημα του πετρελαίου που μας, προμηθεύουν σε εμά και στους Αμερικανούς. Πρόσφατα ε, υπήρξε μια ε, παρατηρήθηκε μια μεγάλη διαφοροποίηση στην ε, προμήθεια του πετρελαίου. Δεν πολλούν μόνο σε εμά και στις Ηνωμένε Πολιτείε. Έχουν πλέον διαφοροποιήσει τους αγοραστές τους και τι αντίκτυπο θα... και αν εξελιχθεί η κατάσταση προς αυτό που ελπίζουμε πίζουμε τον εκδημοκρατισμό, δηλαδή τι συνέπειε θα έχει αυτό για τον παγκόσμιο εφοδιασμό πετρελαίου. Και τέλος, η Ισλαμική απειλή. Ο ρόλος του Ισλάμ. Όπως είπατε και εσεί υπάρχει Ισλαμική τρομοκρατία και η λεγόμενη Ισλαμική απειλή. Μάλλον είναι το μεγαλύτερο θύμα των όσων συμβαίνουν στη Βόρειο Αφρική ή στη Μέση Ανατολή. Ε, γιατί στην, στην πραγματικότητα παραμένουν θεατές των ιστορικών διαδικασιών που εκτελήσονται μπροστά στα μάτια τους και αυτό προκαλεί έκπληξη. Ε, οι ακαδημαϊκοί και οι λεγόμενοι ειδικοί που επί δεκαετίες ε, ετώνιζαν την επιρροή του Ισλάμ έσφαλαν λοιπόν. Εσείς πώς, από πού πιστεύετε ότι εκπηγάζει η νέα απειλή. Ευχαριστώ κύριε Αρλάκη. Κύριε Μέιερ για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καθηγητά Αγγέργε, στην αρχή της παρέμβασής σας είπατε ότι είχαμε υποτιμήσει το πόσο κατεπίγουσα ήταν η κατάσταση της αλλαγής στις αραβικές χώρες. Αυτό κατάλαβα από αυτά που είπε και είπατε ότι είχαμε υποτιμήσει το πόσο επίγουσα ήταν ανάγκη αλλαγής στα αραβικά κράτη. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν θέμα ε, λανθασμένης εκτίμησης. Είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αλλού. Ήταν αλλού και είναι ακόμα αλλού. Το κύριο πράγμα που απασχολεί την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το, η ελευθερία του εμπορίου. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι σε δεύτερη, σε δεύτερη μοίρα. Στην τελευταία παρουσία, στην τελευταία ε, εμφάνιση του κυρίου Κούπερ που είναι ο ειδικό απεσταλμένος Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης στον Μπαχρέιν ο κ. Κούπ πήρε μια θέση η οποία ήταν ίσων αποστάσεων έναντι της κυβέρνησης και των αντιπολιτεύσεων, των αντιπολεμωμένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κατεδίκασε μέχρι και την κατάληψη ενός νοσοκομείου στον Παχρέν από την αντιπολίτευση. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καν μια συγκεκριμένη προσδοκία. Μήπως θα έπρεπε να έχουμε όμως μια διπλωματική στάση πολύ πιο φιλόδοξη. Μήπως θα έπρεπε εμείς να παίξουμε ένα ηγετικό ρόλο σε διπλωματικό επίπεδο και να ξεκινήσουμε από μια διεκδίκηση που να σημαίνει ότι δεν θα έχουμε μια, ένα διπλό πολιτικό λόγο. Άλλο για τις χώρες που έχουν πετρέλαιο και τις χρειαζόμαστε και άλλο για τις χώρες που δεν έχουν πετρέλαιο και δεν εξαρτιόμαστε από αυτές. Παραδείγματο χάρη η Σαουδαραβική δυναστεία, μια από τις πιο αιμοσταγείς και σκληρέ δυναστείε σε όλο τον κόσμο, με σωματικές ποινέ που έχουν καταδικαστεί από την Ηνωμένη αλλά παραμένουν με μια δράση κατά των γυναικών που υπάρχει ειδική αστυνομία για τις γυναίκες για να ντύνονται όπως λέει ο τοπικός Ισλαμικός νόμος. Μια γυναίκα δεν μπορεί να μπαίνει σε δημόσιες κοινωνίες χωρίς έναν άντρα δίπλα τη και παρόλα αυτά για τη Σαουδική Αραβία ποιος ασχολείται. Ποια είναι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιος ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία. Τίποτα, μηδέν. Τίποτα. Και γιατί. Γιατί εξαρτώμαθα από το πετρέλαιο της Σαουδικής Αραβίας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η εξίσωση είναι μια εξίσωση η οποία δεν μπορεί να συνεχιστεί στο μέλλον. Δεν μπορούμε να ακολουθήσουμε μια τέτοια αντιμετώπιση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απολύτω απούσα. Τι μπορεί να περιμένει το Μπαχρέιν, τι μπορεί να περιμένουν άλλε χώρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή μόνο για εμπορικέ συμφωνίε που καλύπτουν τα προβλήματα τη ενεργειακή μα εξάρτηση. Και κλείνω, κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια εμπορική διαμάχη μεταξύ τη Ισπανία, τη Γαλλία και των Ηνωμένων Πολιτειών για να δουν ποιος θα πουλήσει περισσότερα άρματα μάχης στη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι η συμμετοχή μας σε όλη αυτή τη συζήτηση. Ποιος θα, θα πουλήσει πιο πολλά άρματα μάχης στη Σαουδική Αραβία. Αυτό είναι κάτι το απίστευτο. Θα μπορούσαμε με την ίδια λογική να πουλάμε και στο Καντάφι. Γιατί στη Σαουδική Αραβία. Λοιπόν η θέση μας είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να παραμείνει έτσι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να διατηρηθεί έτσι. Ευχαριστώ. Ο κύριος θα κλείσει την Η κυρία Ντεσάγνα θα κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Άκουσα τις απόψεις και τις γνώμες σας. Έχω τρία σχόλια. Πρώτον, επί της ουσίας, πιστεύετε ότι η διεθνής ε, ε, κοινωνία ε, θα πρέπει να ξαναεπινοήσει το δικαίωμα επέμβασης ή το δικαίωμα παρέμβασης, ε, όπως το ονομάζουμε σήμερα. Από ποια στιγμή καθίσταται ζωτική η χρήση του δικαιώματος παρέμβασης. Θα ήθελα την άποψή σας πάνω σε αυτό το ερώτημα, το οποίο πιστεύω θα προκύπτει όλο και περισσότερο στους επόμενους μήνες και χρόνια. Και πιο, τρία πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Στη Σαουδική Αραβία μιλήσατε για τους νέους, οι οποίοι έχουν τις ίδιες προσδοκίες ε, προς την ελευθερία, όπως και όλοι οι νέοι. Δεν μιλήσατε για τις γυναίκες. Έχετε καθόλου στοιχεία για το κατά πόσο υπάρχουν ε, γυναίκες οι οποίες επίσης επαναστατούν κατά ε, όλων αυτών που τους έχει επιβάλει η Σαουδική Αραβία, ε, κατά του καθεστώτος τους, δεύτερον, στη Συρία. Πραγματικά απορώ ε, με τον ε, Σύριο Πρόεδρο, ε, με τον αυτισμό του. Πιστεύετε ότι είναι επάξιος γιος του πατέρα του, και θα δείξει, θα είναι τόσο στενόμυαλος και αυτός όσο ο πατέρας του και θα επιδεικνύει την ίδια πυγμή ή μήπως ποια είναι μάλλον, ποια είναι η ανάλυση σας πάνω στην πολιτική κατάσταση στη Συρία. Εμένα με έχει εντυπωσιάσει αυτή η κόφευση του Σύριου Προέδρου που δεν ακούει τις απαιτήσεις του λαού του, τις διεκδικήσεις του λαού του. Τρίτον, ποιος πιστεύετε ότι είναι ο ρόλος της Τουρκίας σήμερα και αύριο στον αραβικό κόσμο. Ευχαριστώ κυρία Ντεσάχνα. Οκτώ ερωτήσεις λοιπόν υποβλήθηκαν. Ο καθηγητής ε, Γκέργιας έχει 20 λεπτά για να απαντήσει. Εκτός μικροφώνου. Είπα ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσε οι ερωτήσει και θα έπρεπε να έχουμε μια ώρα για να μπορέσουμε να τι απαντήσουμε όλε. Είναι γενικά κριτικού χαρακτήρα ερωτήσεις. Να ξεκινήσω όμως με το πρώτο ερώτημα και μπορώ στη συνέχεια να επεκταθώ περισσότερο. Νομίζω ότι τα τελευταία 60-70 χρόνια η επιλογή ήταν πάρα πολύ σαφής μεταξύ της σταθερότητας από τη μία πλευρά και όλων των άλλων πραγμάτων. Η οι δύσεις, οι δυνάμει και οι Ευρωπαϊκές και οι Ηνωμένε Πολιτείε, αλλά κυρίως οι Ευρωπαϊκοί, οι Ηνωμένε Πολιτείε από την αρχή του ψυχρού πολέμου έφεσαν στο προσκήνιο τη σταθερότητα, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλα αυτά θυσιάστηκαν στο βωμό της σταθερότητας, σταθερότητα, στενή τη ενία, σε ό,τι αφορά την ε, εξασφάλιση της ροής πετρελαίου. Είμαστε όλοι εξαρτημένοι από το πετρελαίο, όχι μονάχα η κατάρα της Μέσης Ανατολής, είναι η κατάρα όλου του κόσμου. Αυτή η κατάρα έχει κάνει μεγάλη ζημιά, όχι μονάχα στις κοινωνίες αυτές που οδήγησε στην εδραίωση των αυταρχικών και καταπιεστικών καθεστώτων, αλλά και σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο η Δύση αντιμετωπίζει αυτό το τμήμα του κόσμου. <clears throat> Αυτό λοιπόν που έχουν κάνει οι δικτάτορες της Μέσης Ανατολής ήταν σαφές. Προσπάθησαν και αυτοί να χειραγωγήσουν αυτή την επιλογή. Ή εμείς ή οι εξτρεμιστές, οι Ισλαμιστές. Λέγαν στις δυτικές δυνάμεις ή εμάς τα έχετε που είμαστε αυταρχικό καθεστώς αλλά σας δίνουμε σταθερότητα, αλλιώς τα έχετε τους Ισλαμιστές. Αν υπάρχει κάτι το οποίο έγινε πια σαφές από τις πρόσφατες εξηγήσεις, αυτό είναι ότι η επιλογή δεν είναι μεταξύ αυταρχικών καθεστώτων των δικτατόρων από τη μια μεριά και εξτρεμιστών από την άλλη πλευρά, υπάρχει αντίθετα ένα πολύ μεγάλο φάσμα. Έχετε αυτούς που βρίσκονται στο κέντρο του πολιτικού φάσματο. έχετε την κοινωνία των πολιτών, έχετε του αγωνιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορούμε να τα βλέπουμε τα πράγματα αυτά απλοποιητικά, μαύρο, άσπρο, αφηρημένα. Το παράδειγμα αυτό λοιπόν το οποίο κυριάρχησε και στην επιστημονική σκέψη τα τελευταία 60 χρόνια δεν υπάρχει πια. Και έχετε τα δίκιο. Ο κύριος χαμένος από όλη αυτή τη διαδικασία είναι η Αλκάιδα και η ιδεολογία της. Αν σκεφτείτε τι ήταν η ιδεολογία αυτή. Ότι η πολιτική δεν οδηγεί πουθενά. Μόνο η βία και η τρομοκρατία είναι οι τρόποι που μπορεί κανείς να επιφέρει την αλλαγή. Γιατί λέει η Δύση δεν θα επιτρέψει στον αραβικό κόσμο να αλλάξουν τα πράγματα. Μα τώρα έχουμε εκατομμύρια και εκατομμύρια και δεν απλοποιώ. Εκατομμύρια Αράβων και Μουσουλμάνων μίλησαν με μεγάλη σαφήνεια. Η πολιτική έχει σημασία, η κοινωνία των πολιτών έχει σημασία. Έχετε πλήθη που μίλησαν όχι μονάχα ότι και είπαν όχι μονάχα ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η οικονομική κρίση, ότι θέλουν ψωμί. Θέλουν να υπάρχει διαφάνεια στην κυβέρνηση, να υπάρχει διαχωρισμό εξουσιών, θέλουν να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή δημοκρατική στην κοινωνία του. Και από την άποψη αυτή νομίζω ότι πράγματι θα πρέπει να ξανασκεφτούμε το κυρίαρχο παράδειγμα για στι σκέψει για τη Μέση Ανατολή και ιδίω για τη μουσουλμανική Μέση Ανατολή, η επιλογή δεν είναι μονάχα μεταξύ αυτο, ε, αυταρχικών καθεστώτων και Ισλαμιστών. Αλλά είναι πολύ ευρύτερη. Και αυτό είναι ένα από τα κύρια διδάγματα που έχουμε αποκομίσει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι οι Ισλαμιστέ δεν υπάρχουν και δεν θα παίξουν ένα κέριο ρόλο στην κατάσταση αυτή. Αλλά υπάρχουν πολλαπλά πρόσωπα του Ισλαμισμού. Είναι πολυεδρικό το φαινόμενο. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι συντηρητικοί, υπάρχουν οι Ισλαμιστέ οι οποίοι είναι ριζοσπαστικοί και ακόμα και αυτοί που είναι αγωνιστικοί αυτή του είδους της ε, μουσουλμανικής αδελφότητος θα παίξουν ένα σημαντικό ρόλο στην περιοχή αυτή, όχι γιατί είναι η πιο ισχυρή, αλλά είναι η πιο καλά οργανωμένη στο τμήμα αυτού του κόσμου. Αν δούμε τι γίνεται στην ΑΕΤΟ. Πείτε ότι γίνονται εκλογές το Σεπτέμβριο. Οι Ισλαμιστές στην Αίγυπτο θα πάρουν μεταξύ 20 και 30% των ψήφων. Στην Τινησία το ίδιο. Αλλά δεν υπάρχει καμία άλλη πολιτική παράταξη που θα μπορέσει να πάρει 20-30% των ψήφων, γιατί δεν είναι αρκετά οργανωμένη. Και αυτό με φαίνει σε αυτό το οποίο μπορεί να κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να έχουμε <clears throat> τη δυνατότητα τα εκατομμύρια αυτά που ξαναβρήκαν τη φωνή τους να έχουν τη δυνατότητα να οργανωθούν, να δημιουργήσουν κόμματα, να υπάρξει εκ της βάσης μια οργάνωση, θα να έχουν τη δυνατότητα να οργανώσουν σεμινάρια, να μιλήσουν στον κόσμο τα κόμματα αυτά, να έχουν επιρροή στα μέσα ενημέρωσης. Δεν λέω κάτι μονάχα σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο, η διεθνής κοινότητα και όχι μονάχα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βοηθήσουν. Δεν είναι χωρίς καθόλου δύναμη όλοι αυτοί, αλλά χρειάζονται τη βοήθειά μας. Τα τελευταία 45 χρόνια όλοι αυτοί έχουν ζήσει σε μια κατάσταση Η κοινωνία των πολιτών ουσιαστικά δεν υπήρχε υπό το πέλμα του αυταρχικού καθεστώτος. <clears throat> Δεν έχετε λοιπόν τους θεσμού, τους βασικούς επί των οποίων μπορεί να οικοδομήσει κανεί τη δημοκρατία και γι' αυτό χρειάζεται και βραχυπρόθεσμα και μαχικροπρόθεσμα να υπάρξει η βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν θέλω να τρομάξω κανένα. Εγώ δεν φοβάμαι τους Ισλαμιστέ. Οι Ισλαμιστέ, η αδερφότητα μουσουλμάνων, δεν είναι αυτή η κύρια δύναμη στι κοινωνίε τη περιοχή δεν μπορούν να κυριαρχήσουν στις κοινωνίες αυτές γιατί δεν εκπροσωπούν την πλειοψηφία. 70% των Τινησίων ή των Αιγυπτίων ή των πολιτών της Ιεμένης και της Συρίας κτλ. είναι στο κέντρο του πολιτικού φάσματος και θα πρέπει να καταμετρηθεί και η ψήφος τους και η φωνή τους στην, στον πολιτικό χώρο. Όπως είδαμε λοιπόν στην Αίγυπτο, οι Ισλαμιστές είχαν τους μηχανισμούς οργάνωσης για να μπορέσουν να συλλέξουν ψήφους και οι ψήφοι τους μέτρησαν. Αλλά 70% από αυτούς που ψήφισαν τους Ισλαμιστές ήταν, οι 20% ήταν που ψήφισαν οι Ισλαμιστές και 70% είναι αυτοί που είναι του κέντρου, είναι αυτοί που βρίσκονται στο μέσο του πολιτικού φάσματος. Επομένως <clears throat> δεν είναι ο κύριος παράγων πια η Αλκάιντα. Η Αλκάιντα είναι ο κύριος χαμένος από το παιχνίδι αυτό. Και το Ισλάμ το ίδιο δεν είναι η κυρίαρχη δύναμη στην περιοχή αυτή. Επανέρχομαι όμως και πάλι και έρχομαι στο θέμα του, των όπλων και όχι μόνο για τον Καντάφη. Είμαι Αμερικανός παρά το γεγονός ότι ε, διδάσκω στο Λονδίνο. Ο Υπουργός Άμυνας Ρόμπερ Γκέιμς Gates πήγε στη Σαουδική Αραβία πριν από μερικέ μέρε για να καταπραίνει και να καθησυχάσει την κυβέρνηση τη Σαουδική Αραβία ότι η Αμερική είναι ακόμα στο πλευρό του. Και πριν από αυτή την επίσκεψη, το ρωτήσανε αν θα συζητήσετε την εσωτερική κατάσταση τη Σαουδική Αραβίας ή του Μπαχρέν. Και είπε, Όχι, δεν θα συζητάμε τέτοια πράγματα. Την εσωτερική κατάσταση είτε στο Μπαχρέν είτε στη Σαουδική Αραβία γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η σχέση των ΗΠΑ με τον κέριο αυτό εταίρο μας. Ουσιαστικά ο Γκέιτς ήθελε να πουλήσει στη Σαουδική Αραβία τα πιο προωθημένα αντιβαλιστικά συστήματα. Πέραν των 60 δισεκατομμυρίων λοιπόν θα αυτό αυτή η συμφωνία 60 δισεκατομμυρίων ήταν η πιο προωθημένη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Σαουδική Αραβία. Αυτό ήθελε να κάνει λοιπόν, να πουλήσει ένα τέτοιο ε, σύστημα ο Γκέιτς στη Σαουδική Αραβία, αντίστοιχο αυτό που είχαν αγοράσει τα αραβικά ε, Εμμυράτα πριν από λίγους μήνες. Και για να ξανάρθω στην απειλή του Ιράν. Η απειλή από το Ιράν είναι και αυτή μια κρίσιμη απειλή. Δεν θέλω να δημιουργήσω διαμάχες, αλλά φαίνεται, βλέπετε ότι το εμπόριο όπλων είναι μια τεράστια, ένας τεράστιος οικονομικός χώρος. Μετά από όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στην περιοχή, το να μιλάει ο Υπουργός Άμυνας της, ε, των Ηνωμένων να πουλήσει άλλο ένα σύστημα αντιπυραυλικό στην ε, κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας, αυτό δείχνει ποιες είναι οι προτεραιότητες των ΗΠΑ. Το Ιράν δεν είναι μια σημαντική απειλή για τη Σαουδική Αραβία. Ο μόνος κίνδυνος που υπάρχει από το Ιράν είναι ο ιδεολογικός από τους μουλάδες. Σε 125 χρόνια το Ιράν δεν έχει κάνει ε, εισβολή σε κανένα. Υπέστη εισβολή στη δεκαετία του 1980 από το γείτονά, το, Σαμα, το Σαντάμ Χουσέιν. Δεν θέλω λοιπόν εδώ να πω ότι δεν υπάρχει καμιά απειλή από το Ιράν. Πρέπει να το συζητήσουμε το θέμα αυτό. Αλλά στην πραγματικότητα το Ιράν δεν αποτελεί απειλή για τη Σαουδική Αραβία. Είναι το ίδιο πιο τροτό στον ιό της δημοκρατίας από ό,τι άλλες χώρες στην περιοχή αυτή. Μετά από την πτώση του Μουμπάρακ βγήκαν στον δρόμο χιλιάδες Ιρανοί. Είναι μια από τις πιο εξελιγμένες κοινωνίες στην περιοχή. Θυμάστε τι έγινε μετά τις πρόσφατες εκλογές. Το Ιράν προσπαθεί απλώς να αντέξει την θύελα αυτή που έχει ξεσπάσει στην περιοχή αυτή. Πριν από μερικές εβδομάδες, όταν ερωτήθηκε ο Ρόμπερ Γκέιτ σε σχέση με το αν αναμειγνύεται το Ιράν στον Μπαχρέν, είπε όχι, δεν το κάνει, αλλά αν γινόντουσαν πολιτικές μεταρρυθμίσεις θα μπορούσε να παίξει κάποιο ρόλο. Αν δεν γίνουν μεταρρυθμίσεις θα μπορούσε το Ιράν να παίξει κάποιο ρόλο στη συνέχεια. Και αυτό πράγματι μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε όλε αυτέ τι εξελίξει στο Ιράν. Αυτό σιγά σιγά αρχίζει να δείχνει ότι η εστίαση φεύγει από το εσωτερικό επίπεδο σε εξωτερικό επίπεδο γιατί αλλάζουν οι συνθήκες και καταλαβαίνουν και οι Αμερικανοί ότι αρχίζουν να υπάρχουν εκείνοι. Ξέρουν οι αμυντικές βιομηχανίες των Αμερικανών και οι μυστικές υπηρεσίες. Όλα αυτά που ξέραμε από τα, Wiki, τα Wikileaks ξέρουμε ότι το Ιράν δεν είχε παίξει κανένα ρόλο ούτε στην Ιεμένη ούτε στον Μπαχρέν. Θα ήθελε το Ιράν να το κάνει αυτό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε σχέση με αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή το Ιράν προσπαθεί απλώς να επιβιώσει, να διατηρήσει το δικό του καθεστώς και να το προστατεύσει από όλα αυτά που γίνονται στη σύνολη περιοχή. Δεν πιστεύω ότι θα δούμε μια συνταγματική μεταρρύθμιση από την τωρινή απόλυτη μοναρχία που υπάρχει στον πεσικό κόλπο σε συνταγματικές μοναρχίες. Η πραγματικότητα είναι ότι η Σαουδική Αραβία είναι οι ηγέτες των δυνάμεων της αντίδρασης. η Σαουδική Αραβία, και είμαι ομός στο θέμα αυτό, η Σαουδική Αραβία είναι η επικεφαλής των αντεπαναστών στην περιοχή αυτή. Είτε αυτό αφορά την Τινησία, είτε αφορά την ΑΕΤΟ. Έχει παρέμβει ενεργά, όπως είδατε, στον Μπαχρέν. Ανεκδοτικά είναι πάρα πολύ οι, οι σχέσεις του Λιβάνου με τη Σαουδική Αραβία, η Συρία με τη Σαουδική Αραβία βρίσκονται σε μεγάλη ένταση μετά από τη δολοφονία του Αλχαρίζη στο Λίβανο το 2005. Αλλά τώρα βλέπετε ότι ξαφνικά η ηγεσία τη Σαουδική Αραβία κατανοεί αυτά τα οποία γίνονται στην περιοχή ότι είναι πραγματικά μια απειλή για την επιβίωσή τη. Και γι' αυτό έχουν μια κοντινή σχέση με τη Συρία. Ξέρουν οι Σαουδάραβε ότι είναι προ το συμφέρον του να παίξουν ένα ενεργό ρόλο, να μπορέσουν να ξεκινήσουν πολιτικές μεταρρυθμίσεις, να ενισχύσουν, να θέσουν τις βάσεις τουλάχιστον για την κοινωνία των πολιτών, να προσπαθήσουν να προκαταλάβουν οποιαδήποτε εξέγερση γιατί η θύελα αυτή είναι τόσο σημαντική, τόσο ισχυρή, που ακόμα και η ίδια η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να την αντέξει όπως έχουν τώρα τα πράγματα. Και ο, ο ίδιος ο βασιλιάς Σαουδικής Αραβίας πιστεύει ότι όλα αυτά που γίνονται θέτουν σε κίνδυνο την ίδια τους την αντίληψη της τάξης και της σταθερότητας. Και γι' αυτό υπήρξε αυτή η ανησυχία και η ένταση στις σχέσεις ΗΠΑ Σαουδικής Αραβίας τις τελευταίες εβδομάδες και η κυβέρνηση Ομπάμα ε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η σημασία της σχέσης ΗΠΑ Σαουδικής Αραβίας είναι πιο σημαντική από οποιαδήποτε μεταρρύθμιση. Ιστορία και Λιβύη. Θέσατε το ερώτημα του αν η Λιβύη είναι ένα τεχνητό κράτος. Όλη η Μέση Ανατολή είναι ένα κατασκεύασμα. Όπως ξέρετε είναι κάτι το οποίο επινοήθηκε μεταξύ του 1918 και του 1920. Μπορούμε να μιλήσουμε για το Λίβανο, μπορούμε να μιλήσουμε για την Υπεριορδανία, τη Συρία, το Ιράκ. Δεν ξέρω που θα ξεκινήσετε. Πολλοί ανόητοι Αμερικανοί μίλησαν για, το, για τη διάσπαση του Ιράκ σε τρία κράτη. Για μένα ως ε, ακαδημαϊκού και μελετητή της πολιτικής της Μέσης Ανατολής αν υπάρχει κάτι το οποίο είναι σημαντικό να πούμε είναι ότι είναι η πρώτη φορά που στην περιοχή αυτή ο αραβικός λαός προσπαθεί να προσδιορίσει την ίδια του τη μοίρα. Είναι μια στιγμή αυτοδιάθεσης. Ο αραβικός κόσμος ήταν περίπου 500 χρόνια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Στο τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου κατέρευσε η Οθωμανική Αυτοκρατορία και οι απικιακές δυνάμεις ουσιαστικά χώρισαν τις αραβικές χώρες μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας και ακολούθησαν τα μεταπικιακά κράτη όπως αυτά του Μουμπάρακ. Οι άνθρωποι λοιπόν σε αυτές τις περιοχές δεν είχαν ποτέ την αυτοδιάθεση, τη δυνατότητα να καθορίσουν την μοίρα τους. Είναι η πρώτη φορά που εκατομμύρια ανθρώπων λένε πρέπει εμείς να αποφασίσουμε για τη μοίρα μας. Δεν είναι θέμα αμερικανικού εμπεριαλισμού που τους ενοχλεί. Δεν τους ενοχλεί ο εμπεριαλισμός αυτός ή ο ιμπεριαλισμός του Ισραήλ. Μιλάνε για απλά πράγματα, για το ψωμί, για τις θέσεις εργασίας, για διαφάνεια στην κυβέρνηση και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Για μένα αυτό μου θυμίζει την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου. Είναι ο, το τείχος του Βερολίνου για τον αραβικό κόσμο που πέφτει αυτή τη στιγμή. Μπορεί να υπερβάλλω, αλλά βλέπουμε πραγματικά να υπάρχουν σημαντικές ρογμές είναι η αρχή της κατάρρευσης μιας τάξης που βασιζόταν σε αυταρχικά καθεστώτα σε αυτή την περιοχή. Και επομένω αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ιστορικό και επαναστατικό. Ιστορικό γιατί είναι η πρώτη φορά που λαμβάνεται χώρα ε, κοινωνικές επαναστάσεις. Δεν λένε απλώς να διορθώσουμε εδώ και εκεί το σύστημα. Θέλουν να το ρίξουν το σύστημα και να το ξαναφτιάξουν από την αρχή. Η Συρία είναι μια σημαντική περίπτωση. Αυτό που γίνεται στη Συρία μας λέει πάρα πολλά πράγματα έχετε ένα ιδιαίτερα κατασταλτικό καθεστώς και παρόλα αυτά ο κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους, ξέροντας ποιες είναι οι συνέπειες. Ξέρουμε ποιες είναι οι συνέπειες και έχουμε δει κάποιες από αυτές τις συνέπειες, αλλά η πραγματικότητα σας λέει πόσο σημαντική, πόσο εκτεταμένη, πόσο βαθιά είναι η θύελα η οποία <clears throat> έχει ξεσπάσει αυτή την περιοχή. και μου θέσατε το θέμα της ε, φιλελεύθερης παρέμβασης κατά κάποιο τρόπο. Μετά από τον ψυχρό πόλεμο η έννοια της ε, παρέμβασης για την εξασφάλιση της ε, ελευθερίας και της δημοκρατίας έγινε πάρα πολύ δημοφιλής στις ΗΠΑ. Όλο αυτό το παράδειγμα των παρεμβάσεων έχει χάσει την αξιοπιστία του μετά από τον πόλεμο του Ιράκ το 2003, μετά από την παρέμβαση των ΗΠΑ το 2003 που ουσιαστικά ήταν το τελευταίο καρφί στο φέρετρο της, του φιλελεύθερου παρέμβασμού, γιατί ήταν φανερό ότι χειραγωγήθηκε για άλλους λόγους αυτή η αντίληψη. Στην Λιβύη η διεθνής κοινότητα δεν είχε πραγματικά επιλογή γιατί χωρίς την παρέμβαση μπορεί να είχαμε μια πραγματική αιματοχυσία. Αλλά πιστεύω ότι ακόμα και στη Λιβύη η δυτική παρέμβαση κινδυνεύει να παραμορφώσει και να διαφθείρει την εντογενάστη, εντογενάστη δημοκρατική επανάσταση στην Λιβύη. Κατανοώ ότι ορισμένοι μπορεί να θέλουν να υπάρχει μια παρέμβαση αυτού του είδους, αλλά εδώ με σοκάρει όταν βλέπω τους στρατιωτικούς διοικητές να επικρίνουν το ΝΑΤΟ γιατί δεν βομβάτισε περισσότερο. Ουσιαστικά εμπλέκουν το ΝΑΤΟ και τη διεθνή κοινότητα σε μια κατάσταση από την οποία θα δυσκολευτούν να βγουν σε μια κατάσταση η οποία μπορεί απλώς να παρατείνει τη σύγκρουση στη Λιβύη. Θα ήθελα λοιπόν να υπάρχει μια πιο περιορισμένη παρέμβαση. Μια παρέμβαση η οποία θα έχει ανθρωπιστικό και μόνο χαρακτήρα. Που θα είναι νομιμοποιημένη από τα Ηνωμένα Έθνη μέσα σε πάρα πολύ σαφή όρια. Αλλιώς έχετε ένα ηγέτη, έχετε μια ομάδα ηγετών που μπορούν πολύ εύκολα να χειραγωγήσουν αυτή τη σύγκρουση και γι' αυτό ανησυχώ για τη Λιβύη. Γιατί θεωρώ ότι η Δυτική Συμμαχία, όλο και περισσότερο, μπαίνει σε στρατιωτικό επίπεδο, είναι λεγόμενη ολίσθηση της αποστολής, το Mission Creep, και η πραγματικότητα είναι ότι καταρχήν αυτή η παρέμβαση είχε σαν στόχο να προστατεύσει τους άμαχους και όχι να καλύψει ένα κενό εξουσίας, ανεξάρτητα από το τι θα θέλαμε όλοι από εμά. Αλλά δεν είναι αυτή η εντολή που είχε. Και όσο οδυνηρό και να είναι αυτό, και όσο και να θέλαμε να έχει φύγει ο Καντάφη, θα πρέπει να σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο. Γιατί αλλιώς, σε τελική ανάλυση, όλοι θα είμαστε χαμένοι από το αποτέλεσμα αυτό. Η Νομίζω ότι θα ήθελα να δω την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσουν, να υψώσουν τη φωνή τους στη διεθνή κοινότητα ασκώντας πίεση στον Σαλήλ να φύγει. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πραγματικά δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Πρέπει να φύγει. Η, η Εμένη μάλλον θα παραμείνει, θα, θα, μάλλον θα καταρρεύσει εάν παραμείνει στην εξουσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να φωνάξουν σε όλους τους τόνους ότι... και να διεκδικήσουν το δικαίωμα της Ιεμένης στην αυτοδιάθεση. Νομίζω ότι τελείωσε ο χρόνος μου. Σας δώσαμε και κάποιο λεπτό παραπάνω για να σας διευκολύνουμε. Μήπως η πρόεδρος Νίμπλερ θέλει να κάνει κάποια τελικά σχόλια. Okay. Εντάξει, ευχαριστούμε λοιπόν για την παρέμβασή σας. Ιδιαίτερες ευχαριστήσεις στον καθηγητή Γέργες που ήταν τόσο εξαντλητικός, τόσο πλήρης και τόσο προκλητικός πάνω σε συγκεκριμένα ζητήματα. Σας χαιρετώ. Ραντεβού αύριο στις 9 για τη συνέχιση των εργασιών της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Έρεται η συνεδρίαση.